Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, για να σεβαστούμε γενικότερα τις χρονικές προθεσμίες, θα ξεκινήσουμε αμέσως. Ήδη έχουμε κάποια καθυστέρηση. Στο σημείο 13 θα εξετάσουμε τις τροπολογίες όπως προβλέπονται στην έκθεση της κυρίας Βλικεντσίουτε για το Έρασμος, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κατάρτιση, την Εκπαίδευση, την Νεολαία και τον Αθλητισμό. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησης προτείνω να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στον τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος καλύπτει την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της ένδυας βέβαια, όπως και ορισμένους άλλους τομείς, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επαρκώς. Θα μιλήσω πρώτα για την επαγγελματική κατάρτιση και την κατάρτιση των ενηλίκων θα ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δραστήριοι μέχρι τώρα, κατέθεσαν πολλές ενδιαφέρουσες τροπολογίες. Αυτό θα βελτιώσει την νομοδότησή μου και είμαι βέβαια ότι ε, συνεχίζοντας τη συνεργασία θα καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες που θα ενισχύσουν τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Για τους σκιώδεις εισηγητές θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και αυτούς. Ο Μάρτιν Κάσλερ ήταν ιδιαίτερα δραστήριος. Θα ήθελα να το σημειώσω αυτό. Ιταλικά. Ιταλικά kurioje numatyti veiksmai būtų nukreipti. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, προσπαθούμε να το λύσουμε. Šalia veiklaus jaunimo sukurti ir analogišką programą skatinti aktyvumą vyresnių žmonių tarpe. Manau, kad iš tiesų tai yra labai svarbu. Πιστεύουμε lipon, ότι όλα αυτά έχουν σημασία, ιδιαίτερα στην periptosi της προσπάθειας ενθάρρυνσης της ε, λεγόμενης ε, ενεργούς γύρανσης. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα ενισχύσει εν πολύ στη γνωμοδότηση, κάτι το οποίο άλλωστε θα είναι και μια καινοτομία σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα αυτό, όπως είπα, δεν καλύπτει μόνο τους νέους, συνεπώς δεν ενδιαφέρει μόνο τους νέους. Ο κύριος Κάσλερ είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα υπό εισαγωγικά πρόγραμμα, το οποίο θα καλύψει και τους ενήλικους, ακόμα και τους ηλικιωμένους, θα βελτιώσει τις δυνατότητες κινητικότητας των δραστήριων πολιτών τρίτης ηλικίας. Πρόκειται λοιπόν για ένα συνολικότερα νέο πρόγραμμα, αναφέρομαι σε αυτό στο σύνολο της γνωμοδότησής μου. Εμείς θα πρέπει να συγκεντρώσουμε βέβαια την προσοχή μας στο βασικό κομμάτι του περιεχομένου ο τίτλος του προγράμματος δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η τελική απόφαση θα ε, ληφθεί από την Επιτροπή Πολιτισμού. Ε, νομίζω ότι αυτοί προκρίνουν τον τίτλο «Η Ευρώπη των Γενεών». Ενδιαφέρον έχει, αλλά πάντως οι συνάδελφοι τελικά θα πάρουν την τελική απόφαση για τον τίτλο του συγκεκριμένου προγράμματος. Η διαβίου μαθητεία είναι ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο και αυτό ε, θα συμπεριληφθεί. Ε, τώρα η δεύτερη εισηγήτρια έχει κάνει ορισμένες προτάσεις τις οποίες στηρίζω. Αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο άρθρο υπαρίθμων 5 που τίνει στην βελτίωση των συνθήκων ζωής ε, κατηγοριών πολιτών που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα και μάλιστα αφορά και νέους ανθρώπους ηλικιακά. Σε συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές θα επανέλθουμε σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τις εταιρικές συνεργασίες και σχέσεις και που θα πρέπει να ενισχυθούν. Η συνεισηγήτρια, η σκιώδης εισηγήτρια μάλλον, αναφέρεται και στη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά αυτό, την τροπολογία της ε, σκιώδους εισηγήτριας, για να δούμε τι συνέπειες θα έχει. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Στάινμπροκ, όπως ε, και μια άλλη Ιταλίδα συνάδελφο, για τις δικές τους τροπολογίες. Η Ιούτα και άλλοι έχουν προτείνει επίσης και να συμπεριληφθούν και οι ατυπικές μορφές εκπαίδευσης, ιδιαίτερα αυτές οι οποίες καλύπτουν ανάγκες ενηλίκων. Έχουν γίνει προτάσεις μέσω τροπολογιών και σχετικά με τα λεγόμενα κοινωνικά κριτήρια τα οποία θα οδηγήσουν σε επιδοτήσεις σε φοιτητές που δεν θα έχουν αρκετά οικονομικά μέσα στη διάθεσή τους και χρειάζονται χρήματα για να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες κινητικότητας χωρίς ε, να παρεμποδίζονται σε αυτό από την οικονομική τους κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν έτσι ώστε οι φοιτητέ να μπορούν να ταξιδεύουν ευκολότερα, να μπορούν να σπουδάζουν στο εξωτερικό και να συνδυάζουν γιατί όχι την εργασία με την εκπαίδευση για την κατανομή τώρα των μέσων του προϋπολογισμού ανάμεσα στα διαφορετικά προγράμματα. Πολλοί συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες και υποθέτω ότι δεν θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία. Ένας άλλος συνάδελφος έχει προτείνει να βάλουμε μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία το επίπεδο χρηματοδότησης δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο για το σύνολο αυτών των προγραμμάτων από ό,τι είχε δοθεί στην αντίστοιχη περίοδο προγραμματισμού 07 με 13. Αυτές είναι οι βασικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί πάντως. Χρειάζεται σίγουρα να τις επεξεργαστούμε καλύτερα και ελπίζω να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες θα σας παρουσιάσω το συντομότερο δυνατόν. Euh, σας ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε το λόγο. Κάτι να συμπληρώσω μόνο. Αν κατάλαβα καλά, και το θέμα το έχω εξετάσει πολύ λιγότερο επιμελώς από ότι εσείς, αλλά από ό,τι κατάλαβα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η βασική ιδέα είναι να προχωρήσουμε επί τη βάση των επιτυχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των successful stories. Και γι' αυτό αυτό το Εράσμος για όλους ήταν κάτι το οποίο ανταποκρίνεται θα έλεγα σε αυτή την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυτή την εικόνα την οποία επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ενός προγράμματος το οποίο έχει δουλέψει καλά. Τώρα για τα επιμέρους προγράμματα Λεωνάρντο και τα λοιπά και πόσο είναι επί τη χέστερα ή όχι αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί είναι σαφές ότι το βασικό πρόγραμμα το οποίο δούλεψε και φαίνεται ότι δούλεψε είναι το έρασμος. Και εγώ ε, έδειχνα μια κάποια κατανόηση για το πρόγραμμα έρασμος για όλους. Πρέπει να πω ότι είχα προσκαλέσει την αρμόδια επίτροπο να έρθει εδώ έτσι ώστε να παρουσιάσει την πρότασή της και εκφράζω τη λύπη μου γιατί δεν στάθηκε δυνατό να έρθει εδώ. Εμείς κάναμε επανειλημμένα διαβήματα, κάναμε πολλές προτάσεις και νομίζω ότι δεν ήταν σωστό εκ μέρους της απέναντι σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει μια σημαντική αρμοδιότητα κάτι το οποίο φαίνεται άλλωστε και μέσω της δικής σας εκθέσεως. Λυπάμαι πολύ λοιπόν για αυτή την απουσία του πνεύματος συνεργασίας, το σημειώνω και για να το πούμε πιο ευγενικά ε, υπήρξε μια τεράστια δυσκολία να συμβιβαστούν οι διαφορές στον χρονισμό και στις υποχρεώσεις ανάμεσα σε εμά και την Επιτροπή. Πάντως εγώ είδα ένα τίτλο να κυκλοφορεί στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η λέξη Εράσμους. νομίζω ότι αυτό ήταν μια σημαντική απώλεια αν πράγματι επαληθευτεί. Ε, καταλαβαίνω βέβαια ότι όλοι που έχουν τα μικρά τους προγράμματα και τις δικές τους αν θέλετε ιδέες θέλουν να τις προωθήσουν ο καθένας στο δικό του κομμάτι αλλά επειδή το Εράσμου συνολικά είναι κάτι το οποίο έχει πετύχει ε, θα έπρεπε να το προωθήσουμε. Βέβαια κατανοώ την επιφυλακτικότητά σας όταν λέτε ότι κοιτάξτε αυτό δεν είναι τελικά σοβαρό θέμα και ας αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Αρμόδια Επιτροπή. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα συνεχίσω, καταλάβατε τι έχω στο νου μου. Μου λένε ότι ε, έχουμε εδώ ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, να δω αν τυχόν θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος εν τω μεταξύ. Α, ο κύριος Μαν ζήτησε το λόγο. Σε σχέση με αυτά που είπε και η πρόεδρος, το πρόβλημα και ο τίτλος είναι ο τίτλος ε, «Έρασμος για όλους». Έρασμος είναι μόνο για τους ε, φοιτητές. Τι πρέπει να πει για όλους. Έχουμε άλλα προγράμματα, Λεωνάρδος και τα λοιπά για τους άλλους. Έχουμε κοινούς στόχους που θέλουμε να ε, επιτύχουμε στον τομέα της επαγγελματικής ζωή. Υπάρχει, για παράδειγμα, ο χώρος για την ευρωπαϊκή ε, κατάρτιση και διπλώματα. Οπότε, δεν καταλαβαίνω γιατί η αρμόδια επί της Επιτροπής δεν είπε να τροποποιήσουμε τον τίτλο. Λάβαμε πολλά πολιτικά μηνύματα από αυτού. Έχουμε επιτυχημένα προγράμματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ευτυχώς ε, όμως τώρα, ε, εντάξει, παρά το ότι δεν μας αρέσει το πρόγραμμα, ο τίτλος μάλλον, ας το κρατήσουμε. Η Κομισιόν βεβαίως ε, ενδιαφέρεται και συμφωνεί. Όταν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι επιτυχημένο, πρέπει να επιδιώκουμε να παραμείνει επιτυχημένο. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν ε, να δημιουργήσουν πρόγραμμα περιβάλλον ανασφάλειες ενώ είχαμε τόσο ε, επιτυχημένο και ασφαλές περιβάλλον για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Είναι λοιπόν απόλυτα λάθος να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά ίσως να μάθω περισσότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα ήθελα ε, να ακούσω με προσοχή όσα θα υποθούν. Πρόεδρος, ε, όπως βλέπετε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στην Επιτροπή μας. Στον αγαπητό Αντιπρόεδρο θα ήθελα να πω ότι τις ε, επιτυχημένε εμπειρίε πρέπει να τι μοιραζόμαστε με άλλους. Ο κύριος Μπίκα. Ευχαριστώ. Να ε, αναφερθώ σε αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, Τόμας Μαν, με τα οποία συμφωνώ 100%. Αλλά μπορώ να πω αυτό που είπε και η συγγήτρια, ότι σε κάθε περίπτωση η ομάδα μας στην Επιτροπή Πολιτισμού δεν θα ήθελε να αλλάξει ε, το όνομα. Υπάρχουν επιτυχημένα τμήματα. Έρασμος, η νεολαία σε δράση και όλα αυτά. Θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία από αυτού. Οπότε έχουμε τους ίδιους στόχους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντουπάλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε λίγα λόγια να, για να εξηγήσω το όνομα γιατί φαίνεται ότι δημιουργεί πολύ ενδιαφέρον. Ήδη έχει ζητηθεί και στην Επιτροπή Πολιτισμού η γνώμη της Επιτροπής. Οι περισσότεροι έχουν εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που διαπιστώσαμε, έχουμε το πρόγραμμα διαβίου Μάθηση, ένα μόνο πρόγραμμα, με μια, με μια σειρά υποπρογράμματα, όπως το έρασμος και άλλα, αλλά τα άλλα δεν τα ξέρει το κοινό. κανείς ε, ε, από τους φοιτητές ε, που έχουν λάβει κάποια επιδότηση δεν ξέρει το κομίνιος και το Γκρούντβιχ. Δεν ξέρει ότι είναι μέσω της διαβίου μάθησης που έλαβε την επιδότηση και όχι μέσω του έρασμος. Δηλαδή, με βάση την αποτίμηση που έχουμε κάνει, την αποτίμηση επιπτώσεων, θα ήταν πολύ θετικό να αξιοποιήσουμε αυτή την παρουσία που έχει το έρασμος που συνδέεται με την κινητικότητα και τη συνεργασία. Νομίζω ότι το κοινό καταλαβαίνει ότι μπορεί να καλύψει το πρόγραμμα αυτό όλα τα επίπεδα εκπαίδευση. Γιατί τον έρασμο όλοι το ξέρουν. Καταλαβαίνουν ότι συνδέεται με την κινητικότητα και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Αν, μιλήσουμε για τον Γκρούντβιχ, δυστυχώ ελάχιστα άτομα γνωρίζουν περί τίνο πρόκειται. Νομίζω λοιπόν ότι είναι η σωστή επιλογή να προτείνουμε ένα ενιαίο όνομα για ένα ε, πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης με ένα ενιαίο λοιπόν τρόπο. Τα συμπεριλαμβάνει όλα. Αξιοποιούμε λοιπόν ε, τα κέρδη που έχουμε ήδη από την μεγάλη ορατότητα της μάρκας Έρασμος. Οι διάφοροι τώρα τομείς εκπαίδευσης. Να καταστεί σαφές ότι στόχος μας είναι να καλύψουμε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και την νεότητα γενικότερα και εκτεταμένα. Δεν θέλουμε λοιπόν να ευνοήσουμε κάποιον συγκεκριμένο κλάδο στον εκπαιδευτικό τομέα. Βεβαίως ε, θα ε, δώσουμε μεγάλη σημασία και στον ε, τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Αλλά και από τη συζήτηση για την νομική βάση είναι σαφές αυτό. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο οι δραστηριότητέ μας, όσα χρηματοδοτούνται από τον έρασμο, δεν επικαλύπτουν τις προσπάθειες που κάνει το Κοινωνικό Ταμείο. Τέλος. Για τα μειονεκτούντα άτομα, τα μη προνομιούχα. Είναι πολύ σοβαρή η προσπάθεια να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε ήδη την εμπειρία μέσω του προγράμματος Νεότητα σε δράση, όπου κάναμε τι αναγκαίε προσπάθειε για να συμπεριλαμβάνονται τα μη προνομιούχα άτομα, τα, άτομα με ειδικέ ανάγκε κτλ. Ευχαριστώ. Η κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ για τις τροπολογίες σας. Πιστεύω ότι οι επιτυχημένες εμπειρίες πρέπει να συνεχίσουν φυσικά να αξιοποιούνται Πιστεύω λοιπόν ότι το πρόγραμμα που θα προτείνουμε στο Κοινοβούλιο θα μπορέσει να ε, τύχει τη συνένεση όλων των συναδέλφων για να διονύσουμε λοιπόν αυτή την επιτυχημένη εμπειρία μας. Όσον αφορά τον τίτλο, το ανέφερε ο κύριος Μαν, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έδωσε επίση τη γνώμη του από αυτού. Εφιστώ την προσοχή σας ότι στο ότι γίνονται συζητήσεις ε, για το θέμα του τίτλου που είναι συχνά υπερβολικά θεωρητικές. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι ο τίτλος, είναι το περιεχόμενο. Πρέπει οπωσδήποτε ε, να έχει πρακτική σημασία η δράση μας. Λέμε ότι οι πολίτες δεν ξέρουν όλα μας τα προγράμματα, αλλά γι' αυτό φταίμε εμείς. Δεν έχουμε σωστή πολιτική ενημέρωσης, επικοινωνίας δεν έχουμε ενημερώσει αρκετά, δεν μιλάμε αρκετά για τις επιτυχημένες εμπειρίες μας, τα επιτυχημένα προγράμματά μας. Ούτως ώστε να είναι όχι μόνο επιτυχημένα, αλλά και γνωστά. Ευχαριστώ. Ελπίζω θα καταλήξω καλές αποφάσεις. Οπότε λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, η ψηφοφορία Συγγνώμη. Θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες στην επόμενη συνεδρίασή μας, στις 8 Δεκάτου, και η ψηφοφορία θα γίνει στις 9 Δεκάτου. Και η Επιτροπή Πολιτισμού θα έχει ένα μήνα για να ε, λάβει υπόψη πλήρως ε, την γνωμοδότησή μα και θα δούμε τι επιφυλάσσει η μοίρα για τον τίτλο αυτής της πρωτοβουλίας της Κομισιόν Καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή εμένει στην άποψή της. Όποιος ε, κάνει μια πρωτοβουλία, βέβαια εμένει στην άποψή του, αλλά και οι νομοθετικές αρχές ε, θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του θέματος. Τώρα ως σημείο 14. Να ε, σας ενημερώσω σύντομα για την αντιπροσωπεία μας στην Κύπρο. 30 και 31 Οκτωβρίου λέει η Πρόεδρος. Εντυπάπεπε, Σέρκας, ε, Σοσιαλιστές, Ινιές Τσούμπερ Γκουε Επιτόπου ήρθε και η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου εκτός ποσόστοσης βέβαια είναι εκεί για να δεχθεί τους συναδέλφους ε, στην πράξη και έπαιξε άψογα το ρόλο μεσολαβητή με τους, διάφορες, με τους διάφορους συνομιλητές μας. Συναντηθήκαμε με την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρία Χαραλάμπους, που την είδατε και τον Ιούλιο βέβαια, εδώ στην Επιτροπή μας, αναφερθήκαμε στη συνάντησή μας με την κυρία Χαραλάμπους για τα θέματα που θα προωθήσει η Κυπριακή Προεδρία ιδιαίτερα οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, την έκθεση Σαρτιέ, στην οποία αναφερθήκαμε χθε. Αναφερθήκαμε και στο θέμα της έκθεσης Γιασλοβίτσκα για τους ε, αποσπόμενους εργαζόμενους. Εντάξει, μπορεί να μην είναι συναρπαστικές οι παρουσιάσεις ε, επισκέψεων, αλλά είναι πολύ δυσάρεστο ε, να μιλάω και να εργάζομαι με τέτοιο θόρυβο. Μπορεί, μπορώ να παρακαλέσω όλους όσους μπαινοβγαίνουν να μην μιλάνε μπαινοβγαίνοντας. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, όπως έλεγα, στα πλαίσια της έκθεσης κυρίας Γιασλοβίτσκα, μιλήσαμε για το θέμα των λεγόμενων επιχειρήσεων γραμματοκιβώτια. Ξέρετε, στην περίπτωση Φλαμόνβιλ βεβαίω, μία από τις επιχειρήσεις ε, που εμπλέκονταν ήταν μία επιχείρηση που είχε τέτοιες δυνατότητες ε, στην Κύπρο, δηλαδή ήταν γραμματοκιβώτιο, και μιλήσαμε και για το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Μιλήσαμε λοιπόν για τις προτάσεις της έκθεσης Γιούτα Στάντρικ για τον τέταρτο πυλώνα του προγράμματος ΨΥ που αφορά τις εγγύσεις για τους νέους. Η υπουργό μας επιβεβαίωσε ότι κατά την άποψή της θα έπρεπε αυτή η εγγύηση για τους νέους να χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Ταμείο. Εμείς ε, υποστηρίξαμε την άποψη ότι το θέμα της εγγύησης για τους νέους ήταν μια νέα κατάσταση. Λόγω των τεράστιων προβλημάτων αυτής της νέας γενιάς που επιχειρεί να εισέλθει στην αγορά εργασίας, οπότε για να είναι και διαφανές το πρόγραμμα και αποτελεσματικό, δεν θα έπρεπε να το μετωπίσουμε ως κάτι το συνηθισμένο στα πλαίσια του κοινωνικού ταμείου, business as usual, αλλά να υπάρξει ένα συγκεκριμένος μηχανισμός που να είναι εύκολη η προσβασιμότητα σε αυτόν για να υπάρξει μια καινοτομία στο κοινωνικό τομέα. Συνοψίζοντας τις συζητήσεις μας, πρέπει να πω ότι δεν μοιάζει να συμμερίζεται το επιχείρημα αυτό η υπουργό, αλλά είχαμε την εντύπωση επίσης ότι ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ήταν πιο δεκτικός προς το επιχείρημα αυτό. Επίσης, ε, συναντήσαμε τον Υπουργό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, τον κύριο Δημοσθένους, όπου αναφερθήκαμε αναλυτικά στις ε, πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές και την έκθεση βεβαίως της κυρίας Μπλίνκεβιτζούτε για το πρόγραμμα Έρασμος για όλους. Στη συνάντηση λοιπόν με τον κύριο Μαυρογιάννη, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπήρξε πολύ επικοδομητικό κλίμα και για την έκθεση Στάνρουκ αλλά και για την ανησυχία μας λόγω του ότι 25% της πολιτικής συνοχής, της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής να μπορεί να δαπανηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Κοινωνική εταίρη τώρα. Στη συνάντηση αναφερθήκαμε πολύ στο θέμα της ελάχιστης αμοιβή, του ελάχιστου μισθού. Πρώτα είδαμε τους ε, εργοδότες, οι οποίοι μας είπαν ότι οι ελάχιστες αποδοχές ενοχλούν, οι ε, ελάχιστη μισθή και μερομίσθια ε, δεν βοηθάνε την ευελιξία της αγοράς εργασίας και δυνατότητα μετακίνηση των εργασομένων ενώ βεβαίως οι εκπρόσωποι των συνδικάτων μας είπαν ότι ήταν πολύ περιορισμένα τα επαγγέλματα όπου υπάρχει ελάχιστος μισθός, άρα δεν έχει καμία επίπτωση στην ε, ελαστικότητα της αγοράς εργασίας. Αυτά είπαμε λοιπόν και κάναμε και μία επίσκεψη στους χώρους, τους συγκεκριμένους. Επισκεφθήκαμε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι υποδειγματικό, απόλυτα. Συναντήσαμε τους υπεύθυνου ενός ε, γραφείου ευρέσεως εργασίας Είδαμε φυσικά το καλύτερο τέτοιο γραφείο στην καρδιά της Λευκοσίας όπου οι Κύπροι ε, που ψάχνουν για δουλειά και που εξαρτούνται από αυτή την υπηρεσία πρώτα απ' όλα κάνουν μια συνάντηση με τον πόλο Ανατολισμού, ούτως ώστε να τους στρέψουν και προς, και προς το ταμείο που τους δίνει το επίδομα ανεργίας. Και τέλος, τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, πήγαμε και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου μιλήσαμε πιο γενικά για την κρίση και την αναγκαιότητα συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων στην προσπάθεια συντονισμού των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Νομίζω ότι ε, σωστά παρουσίασα και πλήρως την επίσκεψή μας, αλλά επειδή και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν στην ε, επίσκεψη είναι παρόντες, αν θέλουν ε, να συμπληρώσουν, να επιμείνουν σε κάποιο θέμα που ίσως ξέχασα, με χαρά να τους δώσω το λόγο. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εύκολο να προσθέσω οτιδήποτε σε αυτήν την αναλυτική παρουσίαση της Προέδρου. Να σημειώσω όμως ένα θέμα που ειλικρινά με εξέπληξε. Η Πρόεδρος ανέφερε ότι οι εργοδότες θεωρούν ότι η ελάχιστη μισθή και μερομίσθια είναι φραγμός και δυσχέρεια. Αλλά ο ελάχιστη, η ελάχιστη αμοιβή είναι περιορισμένη. Ούτω ή άλλως είναι χαμηλά τα ποσά αυτά και δεν είναι η χώρα αυτή η χώρα με χαμηλά ημερομίσθια και αποδοχές. Αυτό που με εξέπληξε είναι ότι στην Κύπρο, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων και την μετανάστευση, ένα θέμα αναφέρθηκε επανειλημμένα. Το θέμα το πώς θα εμποδιστούν οι ξένοι εργαζόμενοι να μεταναστεύσουν στην Κύπρο και πώς θα κρατήσουν τους δικούς τους νέους στην Κύπρο. Υπάρχει λοιπόν πρόθεση να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, να εμποδιστούν. Με εκπλήσει αυτό. Ενώ συζητάμε για ενιαία ε, αγορά εργασίας. Νομίζω ότι αυτό είναι ανησυχητικό, ειλικρινά το λέω. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Η κυρία Τσούμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου, η επίσκεψη που έγινε από την Επιτροπή μας στην Κύπρο είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Είχαμε το feedback σε σχέση με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Ήθελα μόνο να υπογραμμίσω κάτι που κατεμένει σημαντικό. Η Τρόικα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κύπρο εξάλλου είχε πάρα πολύ μεγάλη επιρροή σε σχέση με την αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων. Αυτή τη στιγμή ε, είναι σε διαπραγματεύσεις η Κύπρος με την Τρόικα για να επιτύχει μια οικονομική βοήθεια και νομίζω ότι είναι σκόπιμο να το τονίσουμε και αυτό και θα μπορούσαμε ενδεχομένω να το αναφέρουμε στο ενημερωτικό σημείωμα ότι και τα συνδικάτα αλλά και οι εργοδότες θεωρούν πως ο κοινωνικός διάλογος και η διάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, κυρίως ως προς τις συλλογικέ συμβάσεις, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι σε σχέση με αυτό, δεδομένου το ότι σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποδιαρθρώνουν εργασιακές σχέσεις που έχουν οικοδομηθεί επί σειρά δεκαετιών. Τα συνδικάτα ανέφεραν ρήτα ότι δεν θα επιτρέψουν η αδίποτε παρεμβολή της ε, Τρόικα ε, στις ε, δικές τους εργασίες και στις δικές τους πρακτικές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Τσούμπερ που αναφερθήκατε σε αυτό το σημείο. Ξαναδιαβάζοντας ε, τις σημειώσεις μου συνειδητοποίησα ότι παρέλειψα ένα πολύ σημαντικό σημείο από τις συζητήσεις μας στη Λευκοσία, το θέμα της Τρόικα και της λειτουργίας της. Και το θέμα της επιρροής της σε σχέση με, την, ε, με το κυβερνητικό επιτελείο και τους, ε, τη Βουλή ή και τους κοινωνικούς εταίρους. Μας εξέπληξε και θα συμφωνήσουν νομίζω τα μέλη της Επιτροπής. Όταν ε, μάθαμε λοιπόν ότι ο Υπουργό Δημοσίων Οικονομικών δεν επικοινωνεί με τους υπολείπους ε, υπουργού σε σχέση με τα αιτήματα ενημέρωσης ή αλλά από πλευρά της Τρόικα, δηλαδή δεν υπήρχε ενημέρωση στη Βουλή σε σχέση με τη φύση ε, των απαιτήσεων και των ε, των όσων απαιτεί η Τρόικα και καμία διαβούλευση ε, με τους κοινωνικούς εταίρους. Στις 13 Οκτωβρίου θα γίνει πάλι συνάντηση με την Τρόικα και πρέπει να έχουμε και αυτό κατά νου. Σε σχέση με αυτά που μας είπε η κυρία Μπάουερ, θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Κύπρο σε σχέση με την εκπαίδευση των νέων και την επανομαζόμενη διαρροή εγκεφάλων για τους νέους είναι πάρα πολύ σημαντικό και τονίστηκε αρκούντω στην επίσκεψη. Ένα τελευταίο σημείο που όμω είναι εξίσου σημαντικό είναι το αίτημα των συνδικάτων ε, σχετικά με ε, τη συμμετοχή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στην όλη διαδικασία, κυρίως όταν παρεμβαίνει η Τρόικα για να επιτύχουμε μια νέα ισορροπία ανάμεσα στους διαφόρους παράγοντες που χαρακτηρίζουν την κατάσταση στην Κύπρο. Ιδού λοιπόν αυτή είναι μια νέα πρακτική, γίνεται προφορική παρουσίαση ε, της κάθε επίσκεψης ε, που κάνει η Επιτροπή μας. Επιστεύω ότι είναι πάρα πολύ θετική η πρακτική, διότι σχηματίζουμε έτσι μια πλήρη εικόνα σε σχέση με ένα απλό σημείωμα. Σίγουρα όλοι διαβάζουν αυτά τα σημειώματα, αλλά δεν αποτυπώνονται στο μυαλό του με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε ένα μακρύτατο κατάλογο ψηφοφορίων. Έχετε όλες τις ηλεκτρονικές σα κάρτε. παρακαλώ. Πολύ ωραία, έχετε εισαγάγει ήδη τις κάρτες στα μηχανήματα, όλα λειτουργούν, δεν χρειάζονται τα καν δοκιμές. Ας αρχίσουμε στο σημείο 15 με την ε, έκθεση του κυρίου Μπέκερ, γνωμοδότηση πρωτοβουλίας σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έχουμε voting list εδώ. Παράγραφ 1, compromis 1, qui est pour. Συμβαστική 1. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Παράγραφο 2, συμβαστική ε, ε, ε, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Παράγραφος 3 συμβαστική κάπα και κάπα Α ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν αναφέρθηκα στο ότι υπάρχει και προφορική τροπολογία για τη συμβαστική κάπα. Υπήρξε κάποια ένσταση, υπήρχε κάποια ένσταση μάλλον για τη συμβαστική κάπα, κύριε Σέρκας. Εκτός μικροφώνου Σχόλια από τον κύριο Σέρκας. Αν υπάρχει ένσταση, τι γίνεται, ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε την προφορική και ε, ψηφίζουμε τη συμβαστική κάπα χωρίς την προφορική τροπολογία. πρέπει να ανατρέψετε μέσα στον κατάλογο ψηφοφορίων και φτάνουμε στην παράγραφο 4, συμβαστική L. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια, παράγραφος 6, συμβαστική M. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 103 έχει αποσυρθεί. Και οι υπόλοιπε καταπίπτουν και φτάνουμε στην παράγραφο 7, συμβαστική εν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 109 έχει αποσυρθεί, η 110 καταπίπτει και φτάνουμε τώρα στην παράγραφο 9, συμβαστική όμικρον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 9 έχουμε την τροπολογία 126 του Σφεν Γκίγκολτ υπέρ κατά αποχές επειδή είναι δύσκολο να κοιτάζω περιμετρικά και να εκτιμώ την έκβαση μιας ψηφοφορίας, ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 126 του κυρίου Σφέν Κίγκολτ. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 19 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε για την 127 της κυρίας Τάινρουκ υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Στην παράγραφο 10 Ψηφίζουμε την τροπολογία 130 του κυρίου Σφεν Γκίγκολ σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Μέχρι το performing the contract. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιοι είναι υπέρ της προσθήκης meet criteria of performing the contract. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 11, συμβαστική π, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 139 περίφθη, φτάνουμε στην παράγραφο 14, συμβαστική Q από τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν μάλλον πάλι για την ίδια παράγραφο 14 έχουμε μια δεύτερη συμβαστική τροπολογία η ΑΡ από τέσσερις πολιτικές ομαθεπείς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15 η τροπολογία 153 της κυρίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 154 της κυρίας Τάινρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 155 της κυρίας Μάνερ καταπίπτει ως εκ τούτου και μετά την παράγραφο 15 θα ψηφίσουμε για τη συμβαστική Y τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια η 157 Κίνγκα Κιόνς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για τον υπότιτλο 3, για το υποτμήμα 3 μάλλον, η ε, 158 υπέρ, παρακαλώ, ε, κατά, συγγνώμη, αποχές, εγκρίνεται. Για το 4, η 184, επίσης διαγράφουμε ένα τμήμα εδώ, Νίλσον και Λούδβιξον, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, ηλεκτρονικός έλεγχος, παρακαλώ, για την 184. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ, 21 ψήφι κατά. Ζητώ συγγνώμη, 18 υπέρ, 21 ψήφι κατά, μία απόχη, όντως απορρίπτεται. Παράγραφος 17, 185 της κυρίας Χίρση και 186 της κυρίας Μπέκερ είναι ταυτόσιμες και τη ψηφίζουμε μαζί. Διαγράφουμε τμήματα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Η παράγραφος 17 απορρίπτεται λοιπόν. Φτάνουμε τώρα στο τμήμα 5, η 191, Νίλσον και Λούντβικσον, επίσης διαγράφεται τμήμα κειμένου υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 19, συμβαστική S, τεσσάρων ομάδων υπέρ, παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Euh, Φτάνουμε τώρα. Ζητώ συγγνώμη που διστάζω στο, στην 20 συμβαστική ΤΑΦ υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21 συμβαστική γιου 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η παράγραφος 22 συμβαστική Β τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 23 συμβαστική W τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 23 έχουμε την παράγραφο 1 που προτείνει η Επιτροπή Ήτρε θα πρέπει να ψηφίσουμε το τέλος αυτής της παραγράφου 1 και την υπόλοιπη τροπολογία να έχουμε καλύψει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 5 της Ιδίας Επιτροπής Βιομηχανίας σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα από το Considers μέχρι το Business Activity. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ποιοι είναι υπέρ του δευτέρου τμήματος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Μετά την παράγραφο 23 και πάλι έχουμε μία πρόταση από την ΙΜΚΟ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24. Συμβαστική τροπολογία X 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 24 τη 231 της κυρίας Ρέγνερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 233 και υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 235 Κιόνς υπέρ κατά αποχές Έχω την εντύπωση ότι απορρίπτεται, αλλά αν θέλετε κάνουμε και μία επαλήθευση. Αν το θέλετε, παρακαλώ, 235. Κύριε Έρη, ένα λεπτάκι να ψηφίσουμε. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι γιατί έχει αρχίσει η ψηφοφορία για την 235. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 18, κατά, 20, 18 ε, υπέρ, συγγνώμη, 20 κατά, μία αποχή και η 235 απορρίπτεται. Ο κύριος Έρη. Ευχαριστώ. Ξεχάσαμε να ψηφίσουμε την 234 παρότι είχε απορριφθεί η προηγουμένη, δηλαδή 233. Monsieur, euh, Κύριε Ωρή, για ποια τροπολογία μου μιλάτε ακριβώς. Για την 234, ε, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, εγώ έσφαλα, Πρόεδρε. και το ζήτημα. Πάλι μετά την παράγραφο 24, 238, Κίνκα Κένς, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 24 προτείνεται. Α, συγγνώμη, 238 επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ζητήθηκε επαλήθευση. Πέρας. 18 προς 22 κατά Σαφέστατα απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 24, τροπολογία 239 κατά πίπτη και φτάνουμε στην παράγραφο 2 της Ήτρε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6 της Ιδίας Επιτροπής υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 26. 245 ε, του κυρίου Μπερμάγια για διαγραφή κειμένου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 246 του κυρίου Μπέκερ υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η παράγραφος 27, συμβαστική Z και Zα, ε, τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ των δύο τροπολογιών, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Η συμβαστική 1α, δύο πολιτικών ΑΑ, α δυο πολιτικων ομαδων ε, ε, υπερ κατα αποχες εγκρινεται αλφα. Παραγραφός 30, συμβαστική ΑΒ τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 31, συμβαστική AEC τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 231 έχει αποσυρθεί. Μετά την παράγραφο 31 θα ψηφίσουμε για τη 282 του κυρίου Γκίγκολτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παραγραφό 31 έχουμε την τροπολογία που καταπίπτει και θα ψηφίσουμε την παραγραφό 9 της Ήτρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 της Ήτρε πάλι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 της ίδιας επιτροπής υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Φτάνουμε στα εκτιμώντα στη τηλεογική σκέψη, Το α, συμβαστική α, τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το εκτιμώντας α έχουμε δύο συμβαστικές β και β α τεσσάρων ομάδων μαζί παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εκτιμώντας ε, σ τροπολογία 20 των ε, Βεργιά Τόγια και Νεντέλτσεβα καταπίπτει. Θα ψηφίσουμε για το εκτιμώντας ε, δέλτα τη συμβαστική ΣΥ τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας ε συμβαστική D ε, τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη F συμβαστική ε τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το εκτιμώντα F, τροπολογία 38 της κυρίας Ρέγνερ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, εκτιμώντας G, συμβαστική F, τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας H, συμβαστική G, τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας I συμβαστική H τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα μετά το εκτιμώντας I φτάνουμε στην ε, τροπολογία 51 της κυρίας Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ζητώ συγγνώμη γιατί έχω ξεχάσει μία τροπολογία στην σελίδα 22 του καταλόγου μετά το ε, εκτιμώντας α η τροπολογία 16 King Είναι κατά ο εισηγητής. Ε, ποιοι είναι υπέρ ε, της 16 παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, φτάνουμε ε, στις λοιπές αιτιολογικές σκέψεις. Ε, η τροπολογία 1 δεν γνωρίζω τους συντάξεις, αλλά τους έχω σε άλλο κατάλογο. Oh. Τροπολογία 1 της κυρίας Ρέγνερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της κυρίας Γκιόνης υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ. Είναι της κυρίας Γκιόνης. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 της κυρίας Ρέγκνερ και Χίρσε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση για την τροπολογία υπέρ 4 Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι πέρας. 16 προς 18, 6 αποχές, Όντω απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε όμως τις υπόλοιπες τροπολογίες. Πολύ ωραία. Για όλες τις υπόλοιπες, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνονται. Θα ψηφίσουμε για το σύνολο τώρα της γνωμοδότησης, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. 36 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον συγγητή μας, τον κύριο Μπέκερ. Καταδείξαμε εμπράκτος ότι αν στη δημοκρατία θέλουμε ένα συνενετικό αποτέλεσμα, ενίοτε πρέπει να δείχνουμε υπομονή και να περιμένουν σε εξέλιξη το χρόνο. Το λέω αυτό διότι έχουμε αναβάλει ε, πολλά και σε την ψηφοφορία, αλλά εστέφθη τελικά με μεγάλη επιτυχία το εγχείρημά σα και θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο σημερινή διατάξεω, 16. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα το πρωί πήραμε ένα mail από την κυρία Όμεν Ρόιτεν και θέλει να αποσύρει τις ε, τροπολογίες της 369. So it Θα είναι πιο σύντομη η ψηφοφορία, αν μη τι άλλο. Merci Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Για την έκθεση της κυρίας Birgit Σίπελ για τις δημόσιες προμήθειες. Θέτω σε ψηφοφορία το άρθρο 1, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1, τροπολογία 121 της κυρίας Τούρουνεν. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ, κατά αποχές δεκτή. Α, διακόπτη η πρόεδρος, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας. 18 υπέρ, 22 κατά, την ίδια πλειοψηφία ε, έχουμε πάντοτε. Ε, πρέπει να σα ομολογήσω εδώ το περίμενα γιατί είναι υπέρ η συγγήτρια. Είχα ξεχάσει την περιμετρική θεώρηση της αίθουσα. Λοιπόν, ε, από τον ίδιο συντάκτη, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 123 και 120 γιατί είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνονται. 124 Λούτβιξον υπέρ. Κατά αποχές. Ε, απορρίπτεται. Άρθρο 2. Ε, η 126 της συγήτρία υπέρ. Κατά αποχές θα κάνουμε την επαλήθευση, πάλι το ίδιο θα έχουμε 18 προς 22, αλλά τέλο πάντων το κάνουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσαν όλοι πέρας. Α, 19 προς 21. Απορρίπτεται. 127 Μανέσκου και Κόχμεχριν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, η σημεία 22 του άρθρου 2 Τροπολογία 14 στις ηγήτρες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 128 της κυρίας Χάρκιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 10. 130. Λούντβικσον υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 11. Συμβαστική Β. Τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. και μετά όλη την ομάδα τροπολογιών συμβαστική Β. Φτάνουμε μετά το άρθρο 11 στην 197 του Ρινένε. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται κατόπιν άρθρο 15 συμβαστική C δύο ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 16 παράγραψε 1 υποτμήμα 1 126 χάρκιν υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε την επαλήθευση. 126 επαλήθευση. 126 λέει η πρόεδρος, αλλά είναι 206, διορθώνει. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε 6 προς 31, 3 αποϊχές. σαφέστατα απορρίπτεται, 207 μανέσκου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 208 δεν είναι παραδεκτή άρα άρθρο 17 συμβαστική ΣΑ τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, άρθρο 24 παράγραφος 1 μετά το εδάφιο 3 νέο εδάφιο που προτείνει η συγγήτρια στην τροπολογία 15 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 24 τροπολογία 16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 μετά την παράγραφο 3 έχω την 223 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. στην 29 υπό παράγραφο 3, παράγραφο 3 έχω την 238 κοχμερίν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Στο 40 παράγραφό 1 την 17 της εισηγητρίας, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 40 παράγραφος 1 υπό παράγραφος 2. Amendement 18. Euh, Τροπολογία 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 242 ράπτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όσοι συζητάτε τα προσωπικά σας, παρακαλώ να μην μείνετε άλλο στην αίθουσα αυτή. 2.43 της κυρίας Ράπτη, ποιοι είναι υπέρ. Όχι, έχει καταπέσει, συγγνώμη. Δεν ψηφίζουμε τη 2.43. Ψηφίζουμε τώρα την 2.44 της κυρίας Ράπτη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.45 Μανέσκο Κοχμερίν και είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2.45. Είναι ασυνήθιστος ο συνδυασμός. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται. Κάποιες αλλαγές συμμαχιών δεν αμείβονται όσο θα έπρεπε. Λοιπόν, ΕΣΑΙΑ 246 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 247 Σάρι ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2.48 της Ιδίας ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 της εισηγήτριας ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.49 Σαρίες Αγιά ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.50 250 λοιπόν Μπορούμε να την ψηφίσουμε γιατί έχει γίνει δεκτή η 248 της κυρία Εσταγιά είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 251 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 252 Μπίρκι Τσίπελ ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 41 συμβιβαστική ε ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Άρθρο 43, παράγραφος 1, 263, Μανέσκου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 264, Ισαγιά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43, 265 Μανέσκου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά για μια στιγμή, για μια στιγμή. Να τελειώσουμε λοιπόν τη 2.65. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και θα ελέγξουμε τώρα την 2.64. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 17 υπέρ, 25 κατά, είναι σαφές ότι απορρίπτεται. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γενναιόδορη με τους ηλεκτρονικούς ελέγχους, αλλά κάτι ήξερα. Λοιπόν, στο άρθρο 43, υποπαράγραφος 2, 266, Μανέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 54 παράγραφος 2. Συμβιβαστική F. Δύο ομάδες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Άρθρο 55. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για το F συμβιβαστικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 34 υπέρ, 8 κατά. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Έχετε το λόγο. Διαδικαστικά θα ήθελα να θυμίσω ότι οι βουλευτές είναι αυτοί που ζητούν τον έλεγχο και όχι οι βοηθοί. Έχετε απολύτως δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Δεν μου το ζήτησε βοηθός, αν μου το είχε ζητήσει βοηθός θα είχα κάνει την ίδια παρατήρηση μετά. η βοηθή είναι παρατηρητές, δεν έχουν ούτε τον δυνατότητα να μιλήσουν, να φωνάξουν ή να χειροκροτήσουν. Αλλά είναι καλοδεχούμενοι στην αίθουσα και βοηθούν πάρα πολύ τη δουλειά μας. Λοιπόν, άρθρο 55, παράγραφος 1, υπό παράγραφος 1, σημείο ε, α μικρό, 269, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, ε, 55 παράγραφος 2 συμβιβαστική G τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές δεκτή συμβιβαστική G φτάνουμε τώρα μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 55 στην 26 ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε τώρα στην 275 εισαγιά ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Δεκτή 28 της εισηγητρίας ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.76 της εισηγητρίας και του κυρίου Κοφεράτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Φτάνω τώρα στην 30 της εισηγητρίας πάντα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 31 το ίδιο ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.77 της Ιδίας και του Κοφεράτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.78 της εισηγητρίας ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.79 Στάινροκ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 της κυρίας Σίπελ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.80 της κυρία Ζίπελ και του κυρίου Κοφεράτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 της εισηγήτριας ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. 34 το ίδιο ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. 2.81 της κυρίας Τσούμπερ ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 282 της κυρία Ζίπελ και του κυρίου Κοφεράτη ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 283 της εισηγήτριας ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 286 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 ε, της εισηγητρίας ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική H, ποιοι είναι υπέρ. Δύο πολιτικές ομάδες την καταθέτουν υπέρ, είπα, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέτουμε τώρα σε ψηφοφορία. Α, α, Ηλεκτρονικός έλεγχος. έκανα λάθος, λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, θέτω σε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τέλος της ψηφοφορίας για τη συμβιβαστική H. 34 υπέρ, ή 7 κατά, συγγνώμη, μαζικά δεκτή. Λοιπόν, οι τροπολογίες δηλαδή 287, ε, 366 ε, και 339 καταπίπτουν. Τώρα έχω την 288 της εισηγήτριας που είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 2.89 της εισηγήτριας πάντα υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 2.90 της ιδίας υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 291 της ιδίας υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Στο 66 έχω τη συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές δεκτή η συμβιβαστική I αγγλικά. Έχουμε τώρα στο άρθρο 66 παράγραφος 2 σημείο δέλτα μικρό στην τροπολογία 39 της εισηγήτριας. Έχει καταπέσει η συγκεκριμένη τροπολογία. Διακόπτη διστάζοντας η πρόεδρος. Κυρία Σίπελ, τι πιστεύετε, στον κατάλογο της ψηφοφορίας λέγεται ότι δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε παρά μόνο σαν προσθήκη στη συμβιβαστική ε, αλλά αλλιώς θα καταπέσει. Κοιτάξτε, μετά από τη σοφή γνώμη της κυρία Σίπελ ψηφίζουμε την 39. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στο 66 έχω τώρα την τροπολογία 40 της κυρίας Σίπελ σαν προσθήκη στη συμβιβαστική I. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στο 67 έχω τη συμβιβαστική J. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στο 69 παράγραφος 1 στην εισαγωγή έχω την 46 της εισηγήτριας που είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έχω μετά πάλα στο 69 στο σημείο α μικρό την 319 Hughes ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έχω την 47 της κυρία Ήπελη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έχω την 320 στο άρθρο 69 Παράγραφος 1 σημείο β μικρό της κυρίας Ισαγιά, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1 β μικρό η 48. Τροπολογία 48 της κυρίας Σίπελ και η 321 του κυρίου Χιούζ είναι ταυτόσιμες, τίθενται σε ψηφοφορία, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 σημείο C. Οι τροπολογίες 49 και 322 της εισηγητρίας και του κυρίου Χιούς τίθενται από κοινού σε ψηφοφορία ούσες ταυτόσημες. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται στο 69 παράγραφος 2. Έχουν την 323 Χιούς. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται την 324 τώρα της κυρία Σίπελ και του κυρίου Κοφεράτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 50 της κυρία Σίπελ ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στο άρθρο 69 παράγραφοι 3 με 4 συμβιβαστική L. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή συμβιβαστική L. Μετά α, έχω στο άρθρο 66 την 2.35 ε, ζήπελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στο 70 έχω τη συμβιβαστική M δεκτή στο 71 συμβιβαστική 1 από δύο πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές δεκτή στο 71 την 343 στην παράγραφο 3 Ζήπελ και Κοφεράτη ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 της κυρίας Ζήπελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στο 71 μετά την παράγραφο 3 έχω την τροπολογία 60 της κυρίας Ζήπελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά έρχεται η 347 Ισαγιά υπέρ κατά αποχές Δεκτή. τα 349 της κυρίας Εσαγιά ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Διστάζω λίγο, γι' αυτό θα ελέγξουμε παρακαλώ την 349. Άρχεται η ψηφοφορία για την 349. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. 28 υπέρ 14 κατά μία αποχή πράγματι γίνεται δεκτή. Μετά το 73 έχω τη συμβιβαστική όμικρον. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στο 75 παράγραφος 1 την 350 του Ρούνεν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 351 του Ρούνεν. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 352 του Ρούνεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 354 Μανέσκου Κοχμερίν ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή στο 76 παράγραφος 2 συμβιβαστική πι αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική πι μεταφτάνουμε στην 64 της κυρίας Σίπελ. Κυρία Σίπελ μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδών από το 64 μέχρι το 71. Κυρία Τσούμπερ, θέλετε μία ξεχωριστά. Λοιπόν, οι τρεις πρώτες μόνο μου. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. 64 με 66 κατά αποχές απορρίπτονται. Τώρα περνάμε στην 68. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 69. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ. Εναντίον αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 360 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 361 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 362 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 363 υπέρ, κατά αποχές Εσείς οδηγείτε. Λοιπόν, θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος στην 363. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 20 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται η 363. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Μου επιτρέπετε να ξαναρχίσει η ψηφοφορία. Να υπάρξει έλεγχος επί της πιθανής επανάληψης της ψηφοφορίας. Κύριε Όρη, μπορούμε να ξαναρχίσουμε την ψηφοφορία. Βεβαίω ευχαριστώ λοιπόν. Έχω την αίσθηση ότι εφόσον υπάρχει μία ψήφος διαφορά πάλι θα απορρίπτεται, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείτε να ξαναψηφίσετε. Λοιπόν, θα ξαναψηφίσουμε. Θα δούμε αν θα υπάρξει επαλήθευση. Ποιοι είναι υπέρ της επαλήθευσης. Υπάρχει ένας από τη σοσιαλιστική ομάδα επιπλέον. Τώρα πάλι ένας από τη σοσιαλιστική ομάδα ψήφισε λιγότερος. Πέρα τη ψηφοφορίας. 23 υπέρ του ελέγχου, 20 κατά. Συνεπώς θα επαναληφθεί ουσιαστικά η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 363. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 363. Ψηφίσατε όλοι. Δύο δεν ψήφισαν, τόσο το χειρότερο. Για αυτούς πέρα τη ψηφοφορια 23 υπέρ, 19 κατά. Η 363 της κυρίας Μανέσκου γίνεται δεκτή. Χωρίς μικρόφωνο. Ε, να παρατηρηθεί ότι εδώ ελέγξαμε τρεις φορές, ε, λέει 22 υπέρ, 20 κατά. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Δεν το κάνουμε για όλες τις ψήφους το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, 75 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 363. Ε, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στο 87 έχω τη συμβιβαστική Q αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Έχω την 76 της κυρίας Ήπελ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τη 367 εισαγιά, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 77. Ποιοι είναι υπέρ της κυρίας Ήπελ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 78 της συγγητρίας ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η κυρία Ζίπερ. Μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδών μέχρι και το 373. Μέχρι λοιπόν το 16. Ποιοι είναι υπέρ όλων αυτών των τροπολογιών. Κατά αποχές απορρίπτονται. Στο 16 συμβιβαστική S αγγλικό. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 83 της κυρίας, του κυρίου Λούντιξον υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 1. Τροπολογία 84 Τούρινεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 2. 85 από 4 ομάδες. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Τροπολογία, ε, συμβαστική Ι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Μετά το 5, 4 ε, από κοινού μαζί, όχι, α, όχι μαζί τροπολογία συγγήτρια. Τροπολογία 2 τη συγγήτρια υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 3 συγγήτρια υπέρ. Κατά αποχέ ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 τη συγγήτρια υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 5 τη συγγήτρια υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. Ετολογική σκέψη 11. Συμβαστική Β. Από τρει ομάδε υπέρ. Κατά αποχέ Εγκρίνεται. Τροπολογία 19, τροπολογία 95. Σε αιτιολογική 19, τροπολογία 95. Κάλμπνοχ, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86, Μανέσκου, υπέρ. Είναι ή είναι συμβατή υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική 25. Α, να ελέξουμε την 96 της κυρία... Πολλές επαληθεύσεις. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 20-20 και τρεις αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα, μετά το 25, τροπολογία W, από τρεις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την 27, τροπολογία 98, της κυρίας Μανέσκου και Μερίν υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 28-99 ίδιοι συγκεκριτές υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογία 29 έχουμε την τροπολογία 100 Μακιντάια Κάμπρνοχ όπου έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα χωρίς τις λέξεις από την άλλη πλευρά, τρει τελείε οικονομικά υποφελέ. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματο. Κατά αποχέ. Αυτό το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Ποιοι θέλουν να προσθέσουμε αυτέ τι λέξει που είχαμε αφήσει απ' έξω. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Μετά το 32, 102 υπέρ παρακαλώ. Κατά απόχες εγκρίνεται, 34, σημαστική ήξε, 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, το 38 η τροπολογία 8 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 107 Μανέσκου υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται θέλετε να κάνουμε μια επαλήθευση για την 107 παρακαλώ, έλεγχος. Ψήφισαν όλοι πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντα 40, τροπολογία 108. Κάρμπνο, Μάκινταρ. υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, 109 της εισηγήτρες υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, εκτιμώντα 41. Ε, συμβαστική τροπολογία Z, α, δύο ομάδων υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Εκτιμών 41 ή 11 της εισηγήτρες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκτιμών 43. Τροπολογία 12 της εισηγήτρες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111. Κρίστενσεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112. Μανέσκου. Κοχμερίν υπέρ. Κατά. Αποχές. γκρίνεται. Έλεγχος για την 112. Tout le monde a pu Ψήφισαν όλοι πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 114 καμπνόχ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας 44 τροπολογία 13 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 115 Κρίστανσεν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 116 ίδιου συντάκτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 Μανέσκου Κοχμέριν υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της νομοδότησης παρακαλώ Non, je pense qu'ils sont tout à fait là. Le vote est clos. Πέρας 30 προς 1, 11 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Σίπελ. Et nous avons eu la démonstration de l'impact. Εμπράκτος και πάλι είδαμε τη σημασία των συμβαστικών τροπολογιών όταν είναι περίπλοκο περίπλοκος ο φάκελος. Ε, σημείο 17. φορέ για την ε, γνωμοδότηση της κυρίας ε, Μανέσκου πάλι για τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά μια κλαδική προσέγγιση για τους τομείς του είδα της ενέργειας των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Άρθρο 11, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1, η 64, υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές απορρίπτεται. 65 της κυρίας Τουρινέν για διαγραφή κειμένου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 11 της ηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 66 του κυρίου Χέντελ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 67 του ιδίου υπέρ. Ναι, με προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ενστάσεις. Ε, όχι. 67 λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 68 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 69 ντόιτς υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 70 Τύρινεν υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 71. Τούρνεν υπέρ. Έλεγχος για την 70. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ψήφισαν όλοι πέρας. 36 υπέρ προς 6 κατά, ξεκάθαρα εγκρίνεται. 71 τούρνεν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 της ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 της ιδίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 της ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 της ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 της Ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 της Ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 Α, θα ελέγξουμε το 83 Άρχεται Ψηφίσατε όλοι πέρας 24, 18 εγκρίνεται, 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, ψηφίσαμε την 84. Την 84. Για την 85. Με, με συγχωρείτε. Την 84 ψηφίζαμε. Θέλουμε να ελέγξουμε την 84. Ελέγχουμε την 84. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 7 υπέρ, 35 κατά. Σαφώς το 85 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 86 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 συγκίτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 Καμπνόχ Μακίνταερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 της ε, είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 31 παραγραφός 1 συμβαστική α από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 31, τροπολογία 94, υπέρ, κατά. Κατά ποιοι είναι παρακαλώ. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 της συγκήτριας, υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 19 συγκήτριας, υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 20 συγκήτριας, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 96 Deutsch υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 55 παράγραφος 1 παράγραφος 1 σημείο σε συμβαστική β από, από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 99 Τούρουνεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 τούρουνεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτε 101 πάξας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 ηγήτριες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 ιδίας υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται 26 ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 70, παράγραφος 5, συμβαστική σε από τρεις ομάδες, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104, Χέντελ. Μπορεί να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες 104 έως 109. Όχι, α, 104 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτε. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 ντόιτς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 Χέντελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 Τούρουνεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 Ιδίας υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 117 ιδίας υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 118 ιδίες υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Ιδίας υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 120 Χέντελ υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 121 ιδίου υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 122 ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτω. 123 υπέρ, ε, 2 υπέρ κατά αποχές Κύριε Όρη, τι ψηφίσατε υπέρ εγκρίνεται 123 λοιπόν Κυρία Χίρς, δεν έχουν εκτίσει απόψεις στους 124 Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 είναι συμβατή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 Deutsch υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 126 Händel υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 127 Ιδίου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 128 ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 ιδίου υπέρ κατά θα ελέγξουμε την 129 Handel άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας 19 υπέρ 23 κατά Απορρίπτεται 129, 130, Händel υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 131, οι δύο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 32 εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 133 Κάμπρ Νοχ Α, συγγνώμη, συγγνώμη. 33 της Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 που είναι τροπολογία πάληψης κάπνο μάκιντα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 μπορεί να ψηφιστεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη 2 τροπολογία 37 Handel υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 τύρινεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η σκέψη 4 Χέντελ για ε, απάλληψη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική δέλτα από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ετελογική 543 Τούρουνεν. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μετά το, την ετελογική 5, τροπολογία 44 Χέντελ. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία, ε, 7, τροπολογία 46 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 47 ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 Deutsch υπέρ ψηφίζουμε την 49 Deutsch υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 κλειβέτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τέσσερα εισηγήτρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πέντε ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πενταδύο κάπνοχ μακίνταρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 ιδίων υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 54 τούρουνεν 54 τούρνων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 συγγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 Deutsch υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 Händel υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 εισηγήτρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 Händel υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 εισηγήτριες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 Händel υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 εισηγήτρες υπέρ κατά 9 λέω 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 Κάπρλοχ Μάκιντάρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 εισηγήτριας ναι μπορούμε να την ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 Κάμπρνοκ Μάκιντάιρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 Τούρουνεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε συνολικά το κείμενο ηλεκτρονικός Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. 38 υπέρ, 0 κατά, 4 αποχές. Συγχαίρουμε την εισηγητριά μας. Και τώρα περνάμε στο 18, όπου θα ψηφίσουμε την έκθεση Thomas Mann για τις ε, υπηρεσίες εδάφους σε όλα τα αεροδρόμια στην Ένωση την οποία έχουμε ε, ε, εξετάσει επανειλημμένα. Άρθρο 12... Συγγνώμη, συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια πρόταση απόρριψης της πρότασης της Κομισιόν που υπέβαλε η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Τροπολογία 25. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, η πρόταση της Κομισιόν δεν απορρίπτεται. Ενώ η τροπολογία απόρριψης Καταλάβατε, καταλάβατε. Ωραία. Περάσουμε στη, στο μακρύ κατάλογο ε, τροπολογιών. Πρέπει όταν κανείς προεδρεύει να έχει τη διπλή άρνηση στο μυαλό του. Τροπολογία 43 τώρα. Στο άρθρο 12, στον τίτλο. Στάινμπρουκ, Θέρκας, Κρίστενσεν, Κοτσολίνο. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 12, παράγραφος 1, συμβαστική ΑΑ. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 12, παράγραφος 2, συμβαστική Α. Τρεις ομάδες. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε, άρθρο 12, παράγραφος 2 νέο. Συμβαστική ΑΒ από τρεις ομάδες, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνονται. Άρθρο 12, παράγραφος 3, συμβαστική Β από τρεις πολιτικές ομάδες, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 12, παράγραφος 4. Τροπολογία 6 και 54 που είναι ταυτόσημα, τα ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Καταργείται παράγραφος 4, άρθρο 12, παράγραφος 5, τροπολογία 55, απάλληψης υπέρ που έχει υποβάλει η Σκριζλεύσκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 12, παράγραφος 5. Συμβαστική σε από τρεις ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 12 παράγραφος 6. Τέσσερις ε, ταυτόσιμες ε, απαλλητικές τροπολογίες. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνονται. Άρθρο 12 παράγραφος 7. Τέσσερις απαλλητικές τροπολογίες 9, 60, 62 μαζί υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρο 12, παραγραφός 8, τρεις τροπολογίες απάλληψης, 10, 63, 64, τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Οπότε, άρθρο 12 παράγραφος 9 όπου έχουμε τροπολογία 11, 66 και 67 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρο 12. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 68. Κλειβέτη, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 12, παράγραφος 10, μία νέα παράγραφος τώρα. Τροπολογία 69, κλειβέτη και με μία προφορική τροπολογία. Έχει κανείς αντίρρηση για την προφορική, όχι. Ψηφίζουμε την 69 λοιπόν, όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ της ίδιας κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 20 συμβαστική D από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 34 παράγραφος 1. Συμβαστική ε από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 παράγραφος 2. Τροπολογία 79. Μπένιον Ντεμπάκερ. Τροπολογία απάλληψης. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε τη συμβαστική F από τέσσερις ομάδες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 34. Παράγραφο 3. Συμβαστική Ζ. Για το εισαγωγικό τμήμα από τρει ομάδε υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Υπέρ. Φωντανία υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 16. Του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 Στάινμπρουκ Σέρκας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 εισηγητή υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα κάνουμε έλεγχο. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 21-18. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τροπολογία 20 εισηγητού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 39, παράγραφος 1, σημείο 1, συμβαστική HA από τρεις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 39, παράγραφος 1, σημείο όμικρον. 22-95 ταυτόσημα. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Μετά το τροπολογία 96, Στάιμπρουκ Θέρκας υπέρ. Κατά Αποχές. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ και πάλι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Τροπολογία 23 του υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 40. Συμβαστική H από τρεις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική 17. Συμβαστική I. Τρεις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική 17, τροπολογία 31. Σκριντλεύσκα, υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 32 ιδίας υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική 28, συμβαστική J, 4 ομάδων υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική 28, τροπολογία 37, Κρίστεν Στάινρουκ, υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Αιτιολογική 31 συμβαστική κάπα, τρει ομάδε υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Μετά αιτιολογική 31 τροπολογία 41 Κρίστενσεν υπέρ, κατά απόχε, εγκρίνεται. 42 Χέντελ υπέρ, κατά Ποιοι είναι κατά παρακαλώ. Αποχές απορρίπτεται. Μετά το 1, ένα νέο τμήμα μέσω του συμβασμού τεσσάρων ομάδων. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρώτη φορά βλέπω συμβαστική για μια αιτιολογική αναφορά. Αυτό δείχνει τη δημιουργικότητα και την κοινωνική καινοτομία. Τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά συνολικά το κείμενο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 36 υπέρ 4 κατά. Μία αποχή. Συγχαίρουμε τον εισηγητή μας. Οπότε θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τον εισηγητή μας να υπερασπιστεί όλα αυτά τα σημεία φλογερά στα πλαίσια της Επιτροπής Μεταφορών. Και περνάμε στο 19, όπου θα ψηφίσουμε την έκθεση πρωτοβουλίας. Όχι, την έκθεση. της κυρίας Κίνγκα Γκούνς, γνωμοδότηση για την ΙΜΚΟ, για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 3, τροπολογία 43. Μπεναράμπα του, υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 8, εισηγήτρες υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 9, ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο σημείο B, συμβαστική H, από τέσσερις ομάδες, όχι, τρεις ομάδες, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 5, σημείο, παράγραφος 1, σημείο α, τροπολογία 10, της εισηγήτριας, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I από πέντε ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 7 για το εισαγωγικό τμήμα της παραγράφου 1, συμβαστική J. Τέσσερις ομάδες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13, Η συγκίτρια υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14, ιδίας υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 8, σημείο α, συμβαστική K από τέσσερι ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 8 σημείο F ε, υποσημείο 1 παύλα 1 τροπολογία 16 εισηγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 Μπεναράμπα του υπέρ κατά αποχές η κυρία Ήρσου. Ε, έχει δώσει κατεύθυνση υπέρ. Αλλά μετά δεν ξέρω. Να ελέγξουμε λοιπόν την 51. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 21 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 53 ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 χίρς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 9 παράγραφος 2 σημείο B συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 μπεναράμπα του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 Μπεναραμπατού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 χίρς υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 61-62 ε, ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 20 εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 κλειβέτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο α Συμβαστική μη από τέσσερις ομάδες. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στο σημείο B του ίδιου άρθρου και της ίδιας παραγράφου. Τροπολογία 22. Εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23. ιδίες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24. ιδίες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65. Βεναράμπα του υπέρ κατά αποχές 65 ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ πάλι κατά αποχές απορρίπτεται 66 χείρους υπέρ κατά ποιοι είναι κατά τις 66 αποχές εγκρίνεται 67 μπεναράμπα του συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 εισηγήτρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 εισηγήτρες υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται 27 εισηγήτρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 ιδίας υπέρ και περνάμε Έχουμε 28, ε, έχουμε περάσει τα παραρτήματα. Παράγραφο 1. Υπέρ 28 κατα... εγκρίνεται. Ωραία. τολική σκέψη 1. Συμβαστική Α από τρει ομάδε υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ιτολογική 3. Συμβαστική Β από τέσσερι ομάδε υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ιτολογική 5. Τροπολογία 2. Συγκίτρε υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Αιτιολογική 10 συμβαστική σε από 4 ομάδε υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Αιτιολογική 11 συμβαστική D από 4 ομάδε υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Αιτιολογική 13 συμβαστική ε 4 ομάδε υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Αιτιολογική 17 τροπολογία 17 μπιτζότο υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται αιτιολογική 18, τροπολογία 18, ιδίας υπέρ κατά απόχες. Απορρίπτεται αιτιολογική 20, συμβαστική F. Τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται αιτιολογική 27, συμβαστική G. Τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται μετά την αιτιολογική 30. Τροπολογία 41 Händel σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα χωρίς τις λέξεις μέχρι από τότε μέχρι εκεί, χωρίς αυτό το κομμάτι. Ποιοι είναι υπέρ του να μπει το δεύτερο κομμάτι, υπέρ κατά, αποχές, το δεύτερο τμήμα επίσης εγκρίνεται. Με την τολογική 30, τροπολογία 42 του ιδίου υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε συνολικά το κείμενο, ηλεκτρονικός, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 36 πέρα. 0 κατά. 4 αποχές. Συγχαίρουμε την εισηγήτριά μας. Φτάνουμε τώρα στο 20 της ημερησία διάταξης. Πρόκειται για τη γνωμοδότηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με τιμήσατε ορίζοντας με εισηγήτρια. Λοιπόν, συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές θεκτή, συμβιβαστική 2 συμβιβαστική Β μάλλον, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή, παράγραφος 3, τροπολογία 3 Κορνέλισεν, έχει ζητηθεί εδώ και χωρισμένη ψηφοφορία σε δύο τμήματα λοιπόν. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε τώρα της παραγράφου 3 μέχρι εκεί όπου λέγει ε, τρεις από τις οποίες απαιτούν. Κατά αποχές δεκτό το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ του υπολείπου κειμένου, υπέρ κατά απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 3 έχω την τροπολογία 4 Ζαμπόρσκα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 όρη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 6. Α, επαλήθευση στην τροπολογία 5 όρη. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 16 κατά, 16 υπέρ μάλλον, 24 κατά. Πράγματι έχει απορριφθεί. Παράγραφος 5, τροπολογία 6, όροι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7, κορνέλισεν, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 8 τροπολογία 10 όρη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, περνάμε στην 11 Κορνέλσεν υπέρ κατά. Κοιτάξτε, η, η ίδια ψηφοφορία επαναλαμβάνεται λοιπόν. 11 Κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά την 9 έχω την 13 Ζούμπερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 10 έχω την 14 Τσαμπαόρη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 έχω την 15. Τσούμπερ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πριν ψηφίσουμε την παράγραφο 13, ζητώ συγγνώμη από την κυρία Ζαμπόσκα, θα έπρεπε να ψηφίσουμε την τροπολογία της υπαρίθμου 12 που είναι συμβατή με την 11 που ψηφίσατε. 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 13, συμβιβαστική διαγλικό. αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στη 14 έχω τη συμβιβαστική ή αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Μετά έχω την 19 τσούμπερ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έχω τη συμβιβαστική F από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Μετά έχω την 17, την 21 Ζαμπόσκα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 22 Ζαμπόσκα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 23 της κυρίας Ζαμπόσκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φτάνουμε τώρα στην πρόταση σχεδίου συμφωνίας, διοργανικής συμφωνίας, στην παράγραφο 8, το είναι 24 όροι, είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Φτάνουμε τώρα στην ψηφοφορία 13, στην Παύλα 1 συμβιβαστική G αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτό Παύλα 2 27 τσάμπα όρη ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έγινε δεκτή αλλά θα έχει γίνει δεκτή 27 ναι, χωρίς δισταγμό 28 του κυρίου όρη ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 29. Επί της παραγράφου 17 όρη πάντα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο το σύνολο τώρα του κειμένου. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές. Έτσι λοιπόν ε, ορίσαμε την εντολή μας για την ενδιάμεση έκθεση την οποία θα παρουσιάσει η Επιτροπή Προϋπολογισμών κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του μηνός Νοεμβρίου πριν από το Συμβούλιο Κορυφής της 23ης και 24ης Νοεμβρίου. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 21, όπου είναι η τελευταία ψήφος μας Θα συνεχίσουμε με την ίδια επιμέλεια, συμβιβαστική α από τέσσερις πολιτικές ομάδες. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική β, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Μετά την παράγραφο α φτάνουμε στην συμβιβαστική L, αγγλικό, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Μετά την παράγραφο α λοιπόν. Διακόπτη πρόεδρος. Υπάρχει ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοφοριών. Αντί για παράγραφος εννοούμε αιτιολογικές σκέψεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αντίθετα από ό,τι κάνουμε συνήθως, σας ζητώ λοιπόν αυτά τα εκτιμώντας να τα ψηφίσουμε πρώτα. Δεν δημιουργεί προηγούμενο αυτό, αλλά εδώ μόνο. Λοιπόν, μετά το α ψηφίζουμε την τροπολογία 6 Μάρτιν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 23 υπέρ, 1 κατά, 15 αποχές, δεκτή σαφώς. Τροπολογία 7, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 10 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 12 έχει καταπέσει. Περνάμε στην 13 της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 1, 15. Τσούμπε, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Στον τίτλο 2, τροπολογία 17 Κορνέλης εν υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 2, 16 τσούμπερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 2 έχω την τροπολογία 18 της κυρίας Τσούμπερ, η οποία όμως καταπίπτει, οπότε θέτουμε σε ψηφοφορία στην παράγραφο 3 την τροπολογία 19, η οποία διαγράφει το κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην παράγραφο 3 έχω τη συμβιβαστική C αγγλικό, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Μετά την παράγραφο 3 λοιπόν τώρα, φτάνουμε τη συμβιβαστική εν αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ακολουθεί στην παράγραφο 4 η τροπολογία 25 Τσούμπερ, η οποία και αυτή διαγράφει το προηγούμενο κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, η τροπολογία 25 δεν γίνεται δεκτή. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική M, παράγραφος 4, με μια προφορική τροπολογία της ομάδας των συντηρητικών. Όχι, υπάρχει κάποιος που είναι κατά της προφορικής τροπολογίας, οπότε τίθεται σε ψηφοφορία η συμβιβαστική ως έχει υπέρ, κατά, αποχές, η συμβιβαστική M λοιπόν ως έχει γίνεται δεκτή. Μετά την παράγραφο 4 έχω την 29 μπενιόν είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 30 επίσης υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 31 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 5 έχω την 32 της κυρίας Μακιντάιρ. Α, έχει καταπέσει, συγγνώμη. Οπότε θέλω να θέσω σε ψηφοφορία μετά την παράγραφο 5, την 33 του κυρίου Μπουλνό. δεν έχω εδώ την άποψη της εισηγήτριας, οπότε θέτω σε ψηφοφορία την 33. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν. Η 33 γίνεται δεκτή. Μετά την 34 τώρα του Μπενιό, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στο κεφάλαιο 3 έχω την 36 Κορνέλισεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 6. Συμβιβαστική Αγγλικό που παρουσιάζουν τρεις πολιτικές ομάδες ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στην παράγραφο 7 έχω την κάπα αγγλική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή η συμβιβαστική και η αγγλική. Παράγραφος 7. Την τροπολογία 40. Έχει καταπέσει. Θέτω σε ψηφοφορία λοιπόν μετά την 7 την 41 Μάκιντάρ Κάπνο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ποιοι είναι κατά παρακαλώ. Ποιοι απέχουν. Γίνεται δεκτή. Μετά την παράγραφο 7 Έχω τη συμβιβαστική F που έχει κατατεθεί από τέσσερις πολιτικές ομάδες και είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 8, η 43 Κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά την παράγραφο 8 έχω την 44 Κορνέλισεν ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κοιτάξτε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 44, για την τροπολογία 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 22 υπέρ, 18 κατά. Γίνεται δεκτή. Μετά στην παράγραφο 9 έχω την η αγγλικό συμβιβαστική ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 5. Έχω την 45, έχει καταπέσει όμως. Ψηφίζουμε λοιπόν μετά την 9, την 49 μπενιόν, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Έχω επίσης την 50 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 10, συμβιβαστική G αγγλικό, ποιοι είναι υπέρ Α, λάθος, έχει ζητηθεί εδώ και χωρισμένη ψηφοφορία που κατατέθηκε από το ΕΛΚΑ. Λοιπόν, συμβιβαστική G ως έχει στο σύνολό της, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Και τώρα, τώρα διορθώνει η Πρόεδρος, φτάνουμε στον τίτλο 5, στην τροπολογία 58 Κορνέλισεν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Στην παράγραφο 11 έχω τη συμβιβαστική H αγγλικό από τέσσερις πολιτικές ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στην 11 πάντα έχω την τροπολογία 60, η οποία έχει καταπέσει. Και φτάνουμε μετά την παράγραφο 11 στην τροπολογία 61 Μπουλόν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 62. Τσούμπερ. Θέλετε να υπάρξει έλεγχος για την 61 μπουλάν. Πέρα της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 8 κατά. Γίνεται δεκτή, ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Μπουλά. Στο 62 έχει καταπέσει. Φτάνουμε λοιπόν στην 12, στην 63 τσούμπερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 64. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 12 έχω την 65 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά την παράγραφο 12 έχω την 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στον τίτλο 7 έχω την 67 της ηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Μετά έχω την 68 στην 13. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Μετά την παράγραφο 13 έχω την τροπολογία 69 της κυρίας Κίνγκ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 70 τσούμπερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 ε, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 74. Μπουλόν ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή μετά την παράγραφο 14. Έχω τη συμβιβαστική ή αγγλικό από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές δεκτή. Για τον τίτλο 8 έχω την 78 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στην παράγραφο 15 τώρα έχω την 76. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την 15 έχω τη συμβιβαστική J αγγλικό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μετά την 15 έχω την 80. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 της εισηγητρίας υπέρ κατά αποχές δεκτή μετά την 15 έχω την 82 μπουλόν αν γίνει δεκτή θα θεωρηθεί μια νέα παρά... ως μια νέα παράγραφος 14α μικρό υπέρ κατά αποχές δεκτή μετά την 15 λοιπόν έχω την τροπολογία 83 σε δύο τμήματα. Θέτω στην ψηφοφορία το πρώτο τμήμα χωρίς την λέξη αγγλική narrow. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ποιος θέλει να προσθεθεί η έννοια στενός, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά τώρα την παράγραφο 14. Μετά την 15 μάλλον, διορθώνω. Δεν έχουμε τίποτα για να ψηφίσουμε πλέον. Περνάμε στην 16 λοιπόν της κυρίας Κορνέλισεν. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 17, τροπολογία 86 Κορνέλισεν, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 18. 88 της κυρίας Κορνέλησεν υπέρ κατά αποχές δεκτή. Στη 18 πάντα την 87 Τόμας Μαν συμβατή τίθεται σε ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά την παράγραφο 18 έχω τη συμβιβαστική όμικρον από δύο πολιτικές ομάδες. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα το σύνολο του κειμένου Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για τη συμβιβαστική Ο. Ε, δεν είστε βοηθός, αλλά είστε υπάλληλος πολιτικής ομάδας, έτσι δεν είναι. Δεν άκουσα εσάς, άκουσα κάποιον να φωνάζει από πίσω. Λοιπόν, κάναμε την παρατήρηση που κάναμε για τους βοηθούς, ισχύει και για τους υπαλλήλους των πολιτικών ομάδων. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος. Βέβαια παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία. Συμβιβαστική όμικρον. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 16 υπέρ 20 κατά 0 αποχές ε, δεν γίνεται δεκτή. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα την 89. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα το σύνολο του κειμένου. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 33 υπέρ, 4 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τελειώσαμε εδώ. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικασία για να τελειώσουμε καλά και γρήγορα.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 δεν είναι επειδή τελειώσαμε αυτή τη μακρότατη σειρά ε, ε, ψηφοφοριών ότι ολοκληρώσαμε και την ημερήσια διάταξη. Κάθε άλλο το σημείο, το επόμενο σημείο είναι κέρια ε, σημασία και συνιστά μεγάλη πρόκληση για την Επιτροπή μας. Σας καλώ λοιπόν να μετάσχετε ενεργά στι συζητήσει για αυτό το θέμα. Σημείο 22 θα σας παρουσιάσω τη γνωμοδότηση που θα υποβάλουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ θα πρέπει ε, εσπευσμένα να αποφανθούμε για αυτό το θέμα. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους, αλλά πιστεύω αντιλαμβάνεσαι σε ποιο σημείο είναι σημαντικό να ε, δηλώσουμε παρόντες στη συζήτηση που γίνεται για την ε, στάση που θα τηρήσει το Κοινοβούλιο και τη συμβολή του στι εργασίε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου στα πλαίσια τη έκθεση του κ. Χέρμαν Φανρόμπι προς μια ουσιαστική ε, οικονομική και νομισματική ένωση. Όπως γνωρίζετε ήδη, για την Επιτροπή έκωνη ηγήτρια έχει διοριστεί η κυρία Τάισεν, ε, η οποία έχει συντάξει ε, την έκθεσή της επί τη βάση των τεσσάρων τμήματων, ε, κουτιών, πακέτων, στο θέσουμε όπως θέλετε, που παρουσίασε ο πρόεδρος Φαν Ρόμπεϊ όταν παρουσίασε τον Ιούνιο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ε, νέα του πρόταση. Αυτό σημαίνει πως το σχέδιο έκθεσης ε, της κυρίας Τάισεν απαρτίζεται από το θέμα της ε, Τραπεζικής Ένωσης, ε, της Δημοσιονομικής Ένωσης, της Οικονομικής Ένωσης και της ε, δημοκρατικής διάστασης της διαδικασίας. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα εκδώσει επίσης νομοδότηση για το θέμα αυτό. Ε, έχουμε κάποιους περιορισμούς ε, κάθε φορά που συντάσσουμε απλώς γνωμοδότηση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτείνω κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τη συνέχεια. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω αφενός την κατάσταση από κοινωνικής πλευράς καθώς ε, και τα πολιτικά και νομικά συμφραζόμενα. Θέλετε, γνωρίζετε όλοι την κατάσταση. Γνωρίζετε ότι από τις απαρχές της κρίσης, το 2007 και μετά δηλαδή, τα, ε, όσα έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουμε και το ραντεβού το Δεκέμβρη για την εξέταση του ζητήματος Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης συνοδεύθηκε από μια βαθύτατη οικονομικο-κοινωνικοπολιτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι ορισμένες φορές υποτιμούμε τη σημασία της κρίσης και οφείλουμε να τονίσουμε τη σημασία της διότι Πολλοί συμπολίτε μας ε, θεωρούν ότι πρώτα απ' όλα ασχολούμαστε με τα προβλήματα των τραπεζών και πολύ λιγότερο με τις ε, προτεραιότητες για την ε, καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πολιτικό τραπεδίο χαρακτηρίζεται από την έγκριση στο ίδιο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου ενός αναπτυξιακού συμφώνου θα πρέπει ε, να ε, μεριμνήσουμε ώστε να μην παραμείνει κενό γράμμα αυτό το σύμφωνο, αντίθετα να δημιουργήσει μια νέα δυναμική που ε, θα βρει μια συγκεκριμένη έκφανση, δηλαδή ένα, μια νέα έμφαση που θα αποδώσουμε στο θέμα της απασχόλησης. Θυμάστε όλοι ότι ε, ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι μάλλον είναι παροχημένο το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και την επακόλουθη διένεξη και στη συνέχεια όλοι οι πολιτικοί ηθήνοντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πεισματικά ε, διαψεύουν αυτή τη δήλωση και αντιτάσσουν ότι συνιστά σημαντικό στοιχείο τη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος Μπαρόζη στη διάσκεψη για την απασχόληση για την Ευρώπη που έλαβε χώρα την προπερασμένη εβδομάδα και πάλι απίευθυνε νέα έκκληση για να τονίσει ότι ε, πραγματικά αποτελεί αυτό να πω στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας ε, της Ευρώπης ε, και αυτό σε συνδυασμό με τη διαρκή ε, μείωση των μισθών σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει λύση ανάκαμψης. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τον οδικό χάρτη που παρουσίασε ο πρόεδρος Χέρμαν Φανερόμπη, ε, στον οποίο μόλις αναφέρθηκα, όπου και αυτό έχει σημασία. Δεν αναφέρεται τίποτα ούτε για την απασχόληση ούτε και για την κοινωνική πτυχή του προβλήματος. Όμως, αν εξετάσουμε ακόμη και το πρωτογενές δίκαιο τις συνθήκες, ε, μέσα στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής ε, Ένωσης, ε, όλες οι συνθήκες έχουν ούτως οικοδομηθεί και εξάλλου παρενθετικά να πω ότι το έχει τονίσει επανειλημμένα η Επιτροπή μας και παραπέμπουμε πάντοτε στο άρθρο 121 σχετικά με το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, καθώς και στο άρθρο 148 όπου μπορούμε να βρούμε κάποια στοιχεία για την κοινωνική διάσταση, παρότι δεν μιλάμε τόσο συχνά όταν εξετάζουμε κοινωνικά θέματα για, την οικονομική, για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Πάντως, ε, δίνει την εντύπωση ο δικός χάρτης του κυρίου Φανερωπέν δεν υπάρχει καν το, 100, το άρθρο 148 και ότι ε, η κοινωνική διάσταση δεν θα πρέπει απαραίτητα να ληφθεί υπόψη όταν θέλουμε να ενισχύσουμε τον οικονομικό ε, ή δημοσιονομικό ή ακόμη και τραπεζικό πυλώνα του, της οικονομίας της Ευρώπης. Για αυτό το λόγο σας ε, προτείνω ως προς το περιεχόμενο του οδικού χάρτη του κ. Φαν να ε, προτείνουμε προσθήκη για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής που ενέχει μια σειρά προτάσεων, ε, οι οποίες καταγράφονται σε αυτό το έγγραφο που θα σας μοιράσω. Επίσης, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων αναφέρει ότι έχει ε, ξεκινήσει ένας διάλογος για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει ένα, μια ελάχιστη βάση, όχι ένας ελάχιστος μισθός, ένας ελάχιστος κοινό παρονομαστής κοινωνικού χαρακτήρα σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας ε, και που θα αποτελέσει αντικείμενο κοινή ευρωπαϊκής διαχείρισης. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Πέρα από την πρότασή μας από, για την εγγύηση για τους νέους, και μετά την ψηφοφορία για την έκθεση Steinbrook, πιστεύω ότι αυτή η εγγύηση για τους νέους θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτήν την κοινωνική βάση. Ως προς τα επιδόματα ανεργίας, γνωρίζετε ότι η πρόταση κατατέθηκε από τον κύριο Ντελπλά στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και θα ήθελα να τον προσκαλέσουμε στις μελλοντικέ μας εργασίες. Θα, θα συντονιστούμε με τη γραμματεία για να διαπιστώσουμε αν να τον προσκαλέσουμε, αν και πολύ αμφιβάλλω, ε, πριν την ψηφοφορία της γνωμοδότησής μου, αλλά θα πρέπει εκ του να εξετάσουμε το ζήτημα, διότι έχει καθοριστική σημασία για τις εργασίες της δικής μας Επιτροπής. Ε, αυτή η ιδέα του να διαθέτουμε ένα ευρωπαϊκό εργαλείο σε σχέση με ε, την κοινωνική αλληλεγγύη που πρέπει να καταδείξουμε καθώς και ε, σε σχέση με τα επιδόματα που προορίζονται για τις ε, χώρες της ζώνης ευρώ Θα δούμε λοιπόν πώς, ποια επιρροή έχουν όλα αυτά τα προαναφερθέντα στοιχεία στον κοινωνικό διάλογο. Δεν είναι όμως και το καταλητικότερο σημείο αυτών των διαπραγματεύσεων. Είναι όμως μία πτυχή που ε, θα πρέπει να εξετάσουμε δελεχέστερα. Το δεύτερο κεφάλαιο που θα ήθελα να εξετάσουμε είναι Προφανώς η δημοσιονομική ολοκλήρωση και βλέπω τώρα ότι υπάρχει μία αμφισημία στον τίτλο της έκθεσής μου διότι θα πρέπει να συνηγορήσουμε υπέρ ε, της ολοκλήρωσης ε, της ε, κοινή επιτήρησης στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις επί των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αλλά και ε, επί ε, των δράσεων για δημιουργία νέων θέσεων ε, εργασίας. Νομίζω ότι είναι ρόλος μας να υπενθυμίσουμε τα περί άρθρου 9, γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό δεν χρησιμοποιείται το άρθρο αυτό ε, και ε, ε, σχετικά με την δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρότι πρόκειται για οριζόντια ρήτρα, κάποια φωτεινά μυαλά θεώρησαν ότι αναιρείται αυτό το ενδεχόμενο. Πάντως σήμερα δεν χρησιμοποιείται αυτό το άρθρο 9 για σχετικά ζητήματα. Θα πρέπει πάντως ε, να λάβουμε υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις και ε, να συνειδητοποιήσουμε ως προς την ε, φορολογία ότι έχει μετακυληθεί ε, η φορολογία προς την απασχόληση, αποθαρρύνοντας έτσι τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την τάση. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της φοροδιαφυγής που μειώνει την ικανότητα των κρατών μελών να χρηματοδοτήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και αυτό το στοιχείο ε, είναι εκ των όνου κάνευ και πρέπει να το αναφέρουμε εφόσον ο απότερος στόχος μας είναι η αλληλεγγύη, όπως δηλώνουμε, λοιπόν, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της ζώνης ευρώ θα πρέπει να ενωθούν στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής ε, αντί να επιτρέπουν το ένα στο άλλο να διαπραγματεύονται διμερείς συμφωνίες φοροδιαφυγής. L'intégration euh, économique elle-même. Ως προς ε, την ε, οικονομική ολοκλήρωση αυτή καθεαυτή νομίζω θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και το ρόλο των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση που συνδυάζεται με τα εθνικά μεταρρυθμιστικά ε, προγράμματα και τώρα που ψηφίσαμε την έκθεση της κυρίας Κορνέλισεν διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη ούτε καν ε, δαπάνησαν τα κονδύλια που έχουν ε, διοχετευτεί στα εθνικά αυτά προγράμματα δράσης δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια ένα παράδειγμα κατά τη γνώμη μας και θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε ε, όταν συζητάμε την οικονομική ολοκλήρωση των ε, ε, κρατών της ζώνης ευρώ. Ας περάσω τώρα στο θέμα της, να αναφέρουμε μάλλον και το θέμα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας και στη συνέχεια το φορολογικό ντάμπινγκ, την απόσπαση των εργαζομένων που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού μας μοντέλου. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε κάτι που έχουμε επαναλάβει ε, τους τελευταίους μήνες, ε, το χρονοδιάγραμμα και τις μεθόδους εμπλοκής ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων για το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πιστεύω επίσης ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε περαιτέρω ε, το θέμα της ε, κοινωνίας ε, των πολιτών και των διαφόρων κοινωνικών ενώσεων και εταιριών. Πέρα από τη λογική της επιτήρησης και της επιβολής κυρώσεων που διέπουν τις οικονομικές πολιτικές, θα πρέπει να θυμίσουμε το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής μας, την στρατηγική 2020 και να ζητήσουμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, και όσοι με γνωρίζουν σίγουρα θα με έχουν βαρεθεί γιατί με μεγάλο πείσμα για αυτό το θέμα. Να ζητήσουμε, έλεγα λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει κάποια στοιχεία σύγκρισης για τη δράση των κρατών μελών. Διότι ορισμένοι εξήμων ε, συνηγορούν υπέρ της αφαίρεσης των ε, στρατηγικών επενδύσεων από τον υπολογισμό που γίνεται για το σύμφωνο ε, σταθερότητας. Δεν μιλάμε μόνο για τι επενδύσει αναπτυξιακού χαρακτήρα, αλλά αν θέλουμε να εξετάσουμε τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα σε συνδυασμό με το Σύμφωνο Σταθερότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα κράτη-μέλη για την παιδεία, για την υγεία, για τι υποδομέ του, τι έχουν δαπανίσει Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι αυτή η άσκηση, αλλά είναι ιδιαίτερα ισχνή η συγκρισιμότητα των στοιχείων που μας ε, ε, διοχετεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δεν θα ξαφνιάσω κανέναν αν επανέλθω και επιμείνω σε αυτό το σημείο. Τέλος, και εδώ επιλέξαμε μία light διατύπωση, μία φευγαλαία στην έτσι διατύπωση για την διακυβέρνηση ε, στο εσωτερικό του Eurogroup. Και πάλι θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε ε, η αδίποτη ενίσχυση ε, του ΕΚΟΦΗΝ θα πρέπει να περάσει από ένα διάλογο για τον συντονισμό του ΕΚΟΦΗΝ και του ΕΠΣΚΟ. Ζητώ συγγνώμη ε, που μακρηγόρησα, αλλά ε, προσπάθησα να παρουσιάσω τις βασικές γραμμές της εκθεσής μου, κυρία Μπάουρη και κύριο Σέρκας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση αυτή ε, αντιμετωπίζει σφαιρικά τα θέματα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταστεί σαφής η άποψή μας, να ακουστεί η φωνή μας στη διαδικασία αυτή από την ε, κατάσταση που υπήρχε όταν έκανε την ομιλία του κ. που έχει αλλάξει αρκετά η κατάσταση. Αν δούμε για παράδειγμα τι είπε ο κ. Μπαρόζο την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Η ομιλία Μπαρόζο ήταν διαφορετικού επίπεδου, διαφορετική ποιότητα. Διότι κατέδειξε και τόνισε ε, ότι το κοινωνικό μας μοντέλο πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την ε, διαδικασία επιτήρηση των τραπεζών τα χρηματοπιστωτικά προβλήματα δεν είναι τα μόνα σημαντικά θέματα, δεν είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικά από τα κοινωνικά θέματα. Έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ την ομιλία του. Βεβαίω, ε, η οικονομική κρίση ούτω ή άλλω ε, σε κάποια φάση θα μετατραπεί και σε κοινωνική κρίση. Και να προσθέσω τα εξή. <clears throat> Πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Όσο περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Και ιδιαίτερα για τους νέους. Βεβαίως οι θέσεις αυτές της εργασίας πρέπει να είναι βιώσιμες. να μην είναι τεχνητές. Δηλαδή να μην εξαρτώνται πλήρω από ε, ε επιδοτήσει. Διότι αν εξαρτώνται από επιδότηση θα καταργηθούν μόλις σταματήσει η επιδότηση. Ο τρόπος επίση φορολόγηση τη είναι ένα σημαντικό θέμα, σοβαρό. Το φορολογικό βάρος πρέπει ε, να περάσει στην κατανάλωση, δηλαδή ε, κυρίως να επιβάλλονται καταναλωτικοί φόροι. Αν καταλαβαίνω καλά την πρόεδρό μας, αναφέρθηκε σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα επιδοτήσεων. Και περνώντα τώρα στο θέμα της Κύπρου, ο, ο ελάχιστος μισθός στην Κύπρο είναι υψηλότερο από το μέσο μισθό στη χώρα μου. Οπότε ποιο θα πρέπει να είναι το ελάχιστο επίπεδο, θα πρέπει να είναι το, ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής. Να μην βάλουμε λοιπόν την πάρα πολύ ψηλά. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, στην ουσία ε, δεν εξυπηρετούμε τους στόχους μας. Είναι αντιπαραγωγικό. Και κάτι ακόμη. Στο σημείο 3.12 η πρόεδρός μας τονίζει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί το κοινωνικό dumping. Με αυτό συμφωνώ. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε τρόπους για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιθεωρητών εργασίας διότι το κοινωνικό ντάμπινγκ δεν έχει να κάνει μόνο με τους ε, αποσπασμένους εργαζόμενους. Χαίρομαι που μπορούμε να συζητήσουμε κοινέ εμπειρίες όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων από τη χώρα μου, στο Λουξεμβούργο για παράδειγμα όπου θα έπρεπε αν ελάμβαναν τις ελάχιστες αμοιβές του Λουξεμβούργου θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Επίσης έχω μία ερώτηση. Στα υποεξέταση θέματα είδα ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 24 Σενάτου, ερχόμενη Δευτέρα. Ε, είναι πολύ περιορισμένο το περιθώριο που μας αφήνεται για υποβολή τροπολογιών. Θα μπορούσαμε να επιμηκύνουμε μια-δυο μέρες αυτή την προθεσμία. Να την παρατείνουμε κάπως. Ευχαριστώ. Όπως τα ξέρετε κυρία Πρόεδρε, ε, θα πάμε στη Γαλλία τις επόμενες μέρες για ομάδε εργαζομένων που συνεδριάζουν, οπότε δεν θα έχουμε δυνατότητα να υποβάλουμε τροπολογίες σε αυτή την τόσο σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Θέρκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω ή τα είπατε εσεί ίδια ή ε, τα είπε και η κυρία Βάουερ. Η συγκυρία πολιτικά με βάση την έκθεση Φαντρών είναι τέτοια που πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το μικρό περιθώριο ελπίδας που μας αφήνει ο κ. Φανρόμπουη και η συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθεί να θέσει στα πλαίσια μιας ανανεωμένης κοινωνικής Ευρώπης το κέντρο της προσοχής μας ε, τον κοινωνικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να διαπιστώσω ότι σε όλες τις πολιτικές ομάδες υπάρχει άποψη ότι αν επικεντρωνόμαστε μόνο στην ΟΝΕ δεν επιτυγχάνουμε αυτά που θέλουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν έτσι. Πρέπει σε μια κοινή πλατφόρμα να επιδιώξουμε να συνδυάσουμε την δημοσιονομική και φορολογική πολιτική, την τραπεζική ένωση, αλλά χρειαζόμαστε επίσης και ένα νέο πυλώνα την ε, δημοκρατική φερεγγιότητα. Αλλά λείπει κάτι ακόμη. Πρέπει να υπάρχει και ένας πέμπτος πυλώνας αυτής της ε, πλατφόρμας όπου, που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Να υπάρχουν και οι πολιτικές απασχόλησεις, οι κοινωνικές πολιτικές. Μία λοιπόν συντονισμένη στρατηγική. Αυτό δεν υπάρχει ακόμη. Γι' αυτό σας συγχαίρω κυρία Πρόεδρε για την ταχύτητα με την οποία αξιοποιήσατε αυτή την ευκαιρία για να υποβάλλετε αυτή την γνωμοδότηση στην ΕΚΟΝ με αυτή την ταχύτητα που την απαιτούν οι περιστάσεις. Αλλά χρειάζεται επίσης και σωστή ανάλυση. Ήδη από την πρώτη σελίδα φαίνεται ότι η εργασία που κάνουμε τώρα οδεύει για τη δημιουργία ενός ε, πλαισίου όπου να συνδυάζονται οι οικονομική με την κοινωνική πολιτική, να συνδυάζονται στο ίδιο επίπεδο με το τραπεζικό και δημοσιονομικό τομέα. όταν μιλάμε επίση για τροποποίηση των συνθηκών στην έκθεση φανερών που επίση πρέπει να συμπεριληφθεί και εδώ αυτό, πρέπει να υπάρξει λοιπόν νομοθεσία, πρωτογενή νομοθεσία. Βεβαίω, ε, εμεί το έχουμε πει επανειλημμένα ω Επιτροπή. Γιατί υπάρχει σαφή ανισορροπία μεταξύ ε, τη οικοδόμηση τη οικονομική και τη κοινωνική Ευρώπη. Όχι μόνο δεν επιχειρείται, αλλά τροχοποιείται η κοινωνική οικοδόμηση και αυτό που είπε η κυρία Μπάερ ότι ήρθε η στιγμή το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να μπει στο κέντρο της προσοχής μας όπως η οικονομική τομή. Αυτό είναι μια πρόκληση. Ίσως να είναι σε μεγάλο βαθμό ουτοπική, αλλά χωρίς μια δόση ουτοπίας δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον ορίζοντα προς τον οποίο βαδίζουμε. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να υποβάλω τροπολογία, αλλά μια ιδέα που είναι ιδιαίτερα ακριβή για τους σοσιαλιστές, την επιδιώκουν δηλαδή, δεν θέλουμε να εκλώσουμε την Επιτροπή, αλλά θέλουμε να τη βοηθήσουμε. Κάτι λοιπόν που προέκυψε και από τη ζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουμε μια οικονομική κρίση, έχουμε μια κοινωνική κρίση, αλλά έχουμε και μια πολιτική κρίση τεράστια και δεν θα λύσουμε την οικονομική κρίση αν δεν επιλύσουμε την ουσία της πολιτικής κρίσης. Δεν υπάρχουν πλέον δεσμοί αλληλεγγύης μεταξύ Ευρωπαίων. Υπάρχει απουσία ελπίδας για το μέλλον. Δεν υπάρχει φιλοδοξία από πλευράς των ηγετών της Ένωσης. Και αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω. Σήμερα υπάρχει ουσιαστική ρήξη του κοινωνικού μοντέλου, βάσει του οποίου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργήθηκε η Ευρώπη έχουμε όντως ρήξη του κοινωνικού συμφώνου που προσπάθησε να συμπεριληφθούν όλα τα, νόμο, τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των κεντρικών κρατών, των περιφερειακών κρατών. Αυτή λοιπόν η θεμελιώδης συμφωνία, το θεμελιώδες σύμφωνο καταστρέφεται αυτή τη στιγμή και χωρίς ένα τέτοιο σύμφωνο όχι μόνο το ευρώ δεν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε νέε προοπτικέ οικονομική, ε, δημοσιονομική, φορολογική πολιτική. Δεν μπορεί να υπάρξει νέα πολιτική, δημοκρατική και κοινωνική. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω. Είναι καλό να μιλάμε για ανεργία, καλό να μιλάμε για τα μακροοικονομικά μεγέθη, για τις μαύρες τρύπε, για τις ελλείψεις στο κοινωνικό τομέα. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι η θεμελιώδης βάση κινδυνεύει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να την αποφύγουμε. Έχει λοιπόν διαρριχθεί αυτό το κοινωνικό σύμφωνο, βάση του οποία, όπω είπαν οι πατέρε τη Ευρώπη, ήταν η βάση για την κοινωνική Ευρώπη και για τα κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι. Y Κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι κάτι το θετικό η πρόταση εκθέσεως την οποία μόλις είδαμε. Όλοι έχουμε τον φιλόδοξο στόχο της ολοκλήρωσης της οικονομικής και πολιτικής αγοράς, ε, ένωσης. Είναι δύσκολο να συνδέσει κανείς τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες με τις μακροπρόθεσμες ανάγκες και προσδοκίες. Και στο πλαίσιο αυτό καλό θα είναι να αποφεύγει κανείς ε, να δημιουργεί mm. κάποια εμπόδια ανυπέρβλητα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ αναλυτικά σε αυτά που είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο για το οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοινωνικό πρότυπο είναι εξίσου σημαντικό με τις τράπεζες. Και πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι τράπεζες καλούνται να εξυπηρετήσουν την κοινωνία. Αυτή είναι σαφώς η άποψη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό ανταποκρίνεται και στις ε, πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια των προσπαθειών για τη βελτίωση της ε, διακυβέρνησης στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, να βοηθήσουμε την ανάπτυξη, να βοηθήσουμε την απασχόληση, και στο συγκεκριμένο πεδίο λοιπόν της κοινωνικής ανάπτυξης έχουμε να κάνουμε με σαφέστατο ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να υπογραμμίσω επίσης ότι στο συγκεκριμένο πλαίσιο θέματα όπως η βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων, το θέμα της δυνατότητας μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων είναι όλα θετικά βήματα σε αυτή τη φάση έχουμε κάπως διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το θέμα της συναπόφασης έχει συζητηθεί ανάμεσα σε εσά Πρόεδρε και τον Επίτροπο Ρένα. Δεν ξέρω λοιπόν <clears throat> αν στο παρόν πλαίσιο μπορεί να βρεθεί μια λύση, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προωθήσουμε και στα πλαίσια αυτής της δύσκολης διαδικασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να παράσχει την απαιτούμενη, θα έλεγα, δυνατότητα ελέγχου. Μια μικρή ερώτηση, λέει η Πρόεδρος. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζει τη συζήτηση η οποία θα ξεκινήσει στο τέλος του χρόνου στο Συμβούλιο. Ε, στην ομιλία του ο πρόεδρος Μπαρόσο για την κατάσταση της Ένωσης ε, άνοιξε το δρόμο θα έλεγα για τον διάδοχό του ο οποίος θα πρέπει να οδηγήσει σε μια μεταρρύθμιση. Ε, ποια θα είναι η συνεισφορά και ποιο είναι το επίπεδο προετοιμασίας τελικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιες είναι οι γενικές διευθύνσεις που θα δραστηριοποιηθούν ιδιαίτερα σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης απασχόλησης. Νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ εγώ να αναφερθώ εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης. Το έργο από άλλη Γενική Διεύθυνση. Φυσικά συμμετέχω στις διμερείς επαφές και ο πρόεδρος φυσικά και σε επίπεδο Προεδρίας και σε επίπεδο Κεντρικής Τράπεζας και Eurogroup για την προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Είναι πολύ ενωρίς για μας να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε πολύ συγκεκριμένα πλέον σημεία. Στα θέματα που συζητιούνται μέχρι τώρα η Επιτροπή έχει κάνει κάποιες προτάσεις ε, συγκεκριμένες για την Τραπεζική Ένωση, για έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, κάτι το οποίο στα πλαίσια της παρούσας κρίσης και στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου Κορυφής του Ιουνίου που ζητήθηκε να κοπεί ο δεσμός ανάμεσα στα δημόσια χρέη και τα πιστοτικά ιδρύματα και να απομακρύνουμε έτσι ένας, έναν από τους πιο επικίνδυνους ε, δεσμούς εμπόδια που έχουμε μπροστά μας. Κοιτάξτε, καταλάβαμε τίποτα για το κοινωνικό κομμάτι, ε, για τη Γενική Διεύθυνση ΦΙΝ πάντως και δεν αναφέρομαι σε σας προσωπικά. Καταλαβαίνω που εμπλέκεστε σε τέτοια διαδικασία, αλλά μην μας λέτε ότι τα θέματα της απασχόλησης δεν είναι πρόβλημά σας. Πώς θα συντονίσετε τις προτάσεις σας με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Δεν αρκεί ο πρόεδρός σας να έρχεται εδώ να κάνει μεγάλες δηλώσεις και να λέει ότι το κοινωνικό το κομμάτι επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και από την άλλη να μην μπορείτε να μας πείτε τι θα προτείνετε για τις ανταλλαγές απόψεων με τους υπολείπους ηγέτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από αυτά τα οποία είπατε, θα ήθελα να μάθω πότε περιμένουμε να συναντήσουμε, πότε θα συναντήσουμε τον Επίτροπο Αντόρ. Ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να θέσουμε και στην ε, συνάντηση ε, των συντονιστών. Κοιτάξτε, έχει προβλεφθεί να συναντηθούμε με τον Επίτροπο στο Στρασβούργο στα πλαίσια της ανοιχτής μορφής συντονισμού. Ε, το είχαμε βάλει στις προτεραιότητες του 2013, αλλά θα προσθέσουμε και το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο στη συζήτηση που προηγήθηκε. Γνωρίζω ότι οι προθεσμίες είναι περιορισμένες, αλλά πράγματι το διακύβευμα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μια πρόταση την οποία έχει συμφωνήσει Ολομέλεια στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, με σημείο χρονικό θα έλεγα εκκίνηση τον μήνα Δεκέμβριο. Από ό,τι φαίνεται η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή έχει ήδη αλλάξει ε, προς το πιο γρήγορο το χρονοδιάγραμμά της και εργάζεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα για να μπορέσει να ψηφίσει την πρότασή της στις 15 Οκτωβρίου. Εμείς την δική μας όμως 9 Οκτωβρίου δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ίσως στις 8 να συναντηθούμε με τον κύριο Ντελπλά. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο επηρεάσει τις συμβιβαστικές μας προτάσεις. Πάντως έχει σημασία στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει ήδη εκινήσει να μπορέσουμε να τον συναντήσουμε. και θα έχουμε την δυνατότητα έστω και με μία μέρα επιπλέον 24-25 του μηνός να κάνουμε τις τροπολογίες μας. Είναι δύσκολο να έχουμε κάτι περισσότερο γιατί απαιτείται να προχωρήσουμε στις συμβιβαστικές, στη διατύπωση των συμβιβαστικών που δεν θα γίνει παρά μόνο στις 2 και 3 του μηνός λόγω των χρονικών περιορισμών που έχουμε όλοι. Αυτό που ξέχασα να αναφέρω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ο πλούτος τον οποίο θα προσθέσει η πρόταση της Επιτροπής Απασχόλησης στην έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Είναι κάτι το οποίο σε επίπεδο θα έλεγα συνθήκης ξεπερνάει ε, το άρθρο 9 και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει υποχρεωτικά σε μια μεταρρύθμιση των συνθήκων. Δεν είμαι υπέρ άμεσα κάτι τέτοιο. Αλλά η συζήτηση και για τα τελικά ποσά. Τι μπορούμε να κάνουμε ε, με μια σταθερή θα έλεγα αναφορά στις ε, συνθήκες. Θα είδατε επίσης ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα επαφής με τους τέσσερις ε, Προέδρους ε, ε, αγνοώντας ουσιαστικά το τι έχει γίνει μέχρι τώρα σε επίπεδο κοινοβουλίου στα πλαίσια της δημοσιονομικής κυρίως συνθήκης. Θα σας κρατήσω ενήμερο σχετικά με το πώς αυτά όλα μπορεί να συνδεθούν με τις δικές μας εργασίες. Εφόσον δεν υπάρχει κάτι επιπλέον πάνω στα θέματα αυτά, θα ήθελα να, κατα... να... ορίσουμε λοιπόν προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών στις... στην αγγλική γλώσσα στις 25 Δωδεκάτη Μεσημβρινή. Συζήτηση 8 Οκτωβρίου. Δεν θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε κανονικές τροπολογίες και συμβιβαστικές. Θα τα εξετάσουμε όλα στις 8 για να τα ψηφίσουμε στις 9 και μετά θα πρέπει να προλάβουμε έτσι ώστε να λάβει υπόψη μας η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή τη δική μας άποψη. Φτάνουμε τώρα στο 23 και θα δώσω το λόγο στον κύριο Θέρκας για την έκθεση πρωτοβουλίας του για την ενημέρωση των εργαζομένων προήμη γνώση των αναδιαρθρώσεων. Έχουν κατατεθεί πάρα πολλές ήδη τροπολογίες. Όχι 78 τροπολογίες που είπα, 418. Έχετε το λόγο κύριε Θέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, έχουν υποβληθεί 418 τροπολογίες. Δεν μπορούσα να τις δω όλες μεταφρασμένες, αλλά έχω την ε, εντύπωση την άποψη θα έλεγα ότι το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο και σημαντικό όπως το εξέφρασαν ε, και πολλοί συνάδελφοι όταν κοίταξαν το κείμενο. Και εγώ συμφωνώ ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας είναι περίπλοκη, αλλά και σημαντική. Όλους αυτούς τους μήνες ήρθα σε επαφή με δίκτυα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων που εδώ και 10 χρόνια βοηθάνε το Συμβούλιο, την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα ότι πρέπει να υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί που να μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε την μεγάλη πρόκληση που αποτελούν οι αναδιορθώσεις. Οι αναδιαρθρώσεις στην τεχνολογία και την οικονομία να μην καταλήγουν στην ε, βιομηχανική απερίμωση της Ευρώπης, την καταστροφή των κυρίων ε, οικονομικών δραστηριοτήτων που οι περιφέρειές μας, οι περιοχές μας οικοδόμησαν τα τελευταία 100 χρόνια που αποτελούν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ευρώπης που αναπτύξαμε. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε θα καταλήξουμε σε καταστροφή και σε μετατόπιση των δραστηριοτήτων τα τελευταία τρία χρόνια. Χάσαμε 10% από τους ε, εργαζόμενους στο βιομηχανικό τομέα. Τι θα γίνουμε λοιπόν, μόνο περιοχή τουρισμού και τραπεζικών υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι αυτός ο στόχος μας. Γι' αυτό στην έκθεσή μου κάνω μεγάλη προσπάθεια να επιληθούν τα προβλήματα που κατά πολύ υπερβαίνουν τα όρια των κρατών μας. Όλοι θυγόμεθα, όλοι πληττόμεθα. Άλλοι πριν, άλλοι αργότερα. Τα στοιχεία για την ανεργία που ε, πρόσφατα είδαμε διαπιστώνουν, μάλλον ε, καθιστούν σαφές ότι και χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προβλήματα ανεργίας. Άρα συνολική πρέπει να είναι και αντιμετώπιση. Σοβαρή λοιπόν η πρόκληση, οικονομικά, κοινωνικά, αλλά και στρατηγική πρόκληση από πολιτικής άποψη. Τι ρόλο θα μπορέσει να παίξει δηλαδή στο μέλλον η Ευρώπη συνεργασία μεταξύ των ε, εθνών. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλε αυτέ τι τροπολογίε, 438 λέει ο εισηγητή, που προσπαθούν να βελτιώσουν το κείμενο. Όπω σα είπα, όλου αυτού του μήνε, από τότε που υπέβαλα το πρώτο σχέδιο, με εμπειρογνώμονε, επιτρόπου και τον ίδιο τον πρόεδρο τη Επιτροπή, με την Προεδρία του Συμβουλίου, με τους κοινωνικούς εταίρους, Ο διάλογος με το Business Europe βέβαια ήταν πολύ δυσχερής γιατί πριν ε, μιλήσουν με μένα ήδη είχαν αποφασίσει μια στρατηγική που δεν ε, στοχεύει στην ε, βελτίωση της κατάστασης. Στόχος τους ήταν να μην υπάρξει αυτή η έκθεση. Να μην έχει δηλαδή τη δυνατότητα το κοινοβούλιο μας να παίξει ρόλο σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για την ιστορία της Ευρώπης. Μίλησε επίση με ε, του ευρωπαϊκού οργανισμού, οργανισμούς, ε, κυρίως με τον οργανισμό του Δουβλίνου που έχει μεγάλη πείρα και γι' αυτό εκπώνησα και εγώ κάποιες ε, τροπολογίες αλλά και κάποια προβλήματα στην κατανόηση που δημιουργήσει η έκθεσή μου που θέλω λοιπόν να την τροποποιήσω και πιστεύω ότι και με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχω και καλύτερου συμβιβασμού. Την Πέμπτη λοιπόν θα έχουμε με πρώτη επαφή με του Κιώδης αλλά θα γίνουν και άλλε επαφέ, Όπως είπε και η Πρόεδρος, η ψηφοφορία που πρόκειται να γίνει στις 9 Οκτωβρίου δεν θα γίνει. Θέλουμε λοιπόν να αποτελέσει σημαντική προστιθέμενη αξία το κείμενό μου και με τη βοήθεια τριών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων θέλουμε να μελετήσουμε τα γεγονότα, όχι τις προκαταλήψεις. Τι θα σήμαινε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, τι θα σήμαινε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, τι θα πρέπει να κάνουμε νομοθετικά και εμεί. Το κείμενό μου λοιπόν θα είναι στη διάθεσή σας την επόμενη εβδομάδα και θα παρουσιαστεί στη συνεδρίασή μας στις 9 Οκτωβρίου που προβλέπαμε να, παλιότερα να ψηφίσουμε. Προσπαθούμε λοιπόν ε, σε αυτή την περίοδο χωρίς προκαταλήψεις να αντιμετωπίσουμε το θέμα να μελετήσουμε την τεράστια τεκμηρίωση, την τεράστια πείρα που υπάρχει στην Ευρώπη για το πώς γίνονται οι αναδιαρθρώσεις, πώς προβλέπουμε, προσπαθούμε να προβλέψουμε τις ανάγκες για αλλαγές και πιστεύω ότι όλοι έχουμε τη βούληση, αν υπάρξει μάλλον βούληση από όλου, θα καταλήξουμε εκεί που θα έπρεπε να καταλήξουμε. Η εκθεσή μου έχει δύο τμήματα. Στο δεύτερο τμήμα κάνουμε μια σειρά συστάσει στην Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι θα προκύψουν μεγάλε δυσχέρειε. Σε αυτό το δεύτερο τμήμα προσπαθούμε να δούμε και με τι νομοθετήματα θα προχωρήσουμε. Να δούμε λοιπόν τι θα πρέπει να κάνουμε από όλε τι προοπτικές Χρειαζόμαστε βεβαίω μια οδηγία, ένα νομοθέτημα. Αλλά πρέπει να δούμε και τι άλλε συστάσει μπορούμε να κάνουμε, τι άλλο είδος ήπιου νόμου, για παράδειγμα, κώδικα δεοντολογίας. Φυσικά μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να δούμε ποια θα ήταν τα κατάλληλα μέσα, ούτω ώστε οι αναδιαθρώσει να γίνονται κοινωνικά με πιο υπεύθυνο τρόπο. Χωρί να συζητήσουμε για τη φύση του νομοθετήματο. Και στο πρώτο τμήμα να συζητήσουμε και τη φύση του νομοθετήματος. Τι είδος ε, νομοθέτημα. Βεβαίω πρέπει να είναι ευρωπαϊκό νομοθέτημα. Εγώ νομίζω πως πρέπει να είναι οδηγία, πρέπει να είναι δεσμευτική. Γιατί όλα τα άλλα μέσα ήδη τα έχουμε επιχειρήσει. Νομίζω ότι δεν ε, βοηθάνε παντού οι συστάσεις. Σε κάποιους τομείς βοηθάνε, αλλά όχι παντού. Αλλά λείπει ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα που να καταργεί τις μαύρες τρύπε που υπάρχουν τώρα στην νομοθεσία. Έχουν ως αποτέλεσμα αυτές οι ελλείψεις το να είμαστε ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε διεθνική αναδιάρθρωση. Να περιορίσουμε το θέμα αυτό σε επίπεδο ενό ε, κράτους και επειδή ακριβώς ε, υπάρχουν ελλείψεις στην νομοθεσία, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια οδηγία ακόμη και αν αυτή η οδηγία ε, θέτει ελάχιστες προδιαγραφές και σέβεται πλήρως την επικουρικότητα και τις δυνατότητες που έχουν οι κοινωνικοί εταίροι για να παρέμβουν. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς περισσότερους από τα τελευταία δέκα χρόνια. Δεν θα επανέλθουμε στο σημείο αφετηρίας της πρώτης ε, πράσινης βίβλου πριν από δέκα χρόνια. Δεν χρειάζεται να ξαναβαδίσουμε ένα τομέα απραξίες όπου λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα οι αγορές ε, και οι ε, μέτοχοι θα αποφασίζουν έχω υποβάλει 20 τροπολογίες για τα πιο σημαντικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιστεύω και όταν θα συζητήσουμε και με τους ε, σκιώδες ηγητές θα αναφερθώ στους τροπολογίες των άλλων ομάδων πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεσή μου μεταξύ των εμπειρογνωμών προκάλεσε τέσσερις Αντιδράσει Και για να αντιμετωπίσω αντιδράσει του, υπέβαλε 20 τροπολογίες. Οι ανησυχίες τους και αντιδράσει του έχουν να κάνουν και με τις διαστάσεις τη έκθεσης. Προσπαθώ λοιπόν εγώ να είμαι ε, αρκετά σύντομο και δεν αναφέρω αναλυτικά όλα τα μέσα. Τώρα όμω με τι τροπολογίες πρέπει να ε, είμαι λίγο πιο αναλυτικός για να ε, αντιμετωπίσω κάποιε παρανοήσει και ανησυχίες. Το πρώτο πρόβλημα είναι το πεδίο εφαρμογή. Όπω ξέρετε, θέλω πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογή για το είδος επιχειρήσεων, αλλά πολύ μεγάλο όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων. Μιλάμε για το 1,2% των επιχειρήσεων που έχουν πάνω από 500 εργαζομένους, αλλά αυτοί απασχολούν πάνω από 25% των εργαζομένων, αυτές οι επιχειρήσεις. Μου έγιναν λοιπόν ερωτήσει Γιατί να μην επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή και άλλες αιτήσει που λένε να μην ορίσουμε τον αριθμό των εργαζομένων. Να το συζητήσουμε. Δεν είναι τόσο θεμελιώδες. Αυτό που πρέπει να είναι σαφές είναι ότι είναι μια ελάχιστη προδιαγραφή και η τροπολογία μου 136 λέει ότι αυτό το κατόφλι θα μπορούσε να μειωθεί από την εθνική νομοθεσία ή από συλλογικέ συμβάσει σε κάθε κράτο μέλο. Είναι μια ελάχιστη προδιαγραφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτέ οι 500 θέσει εργασία, 500 εργαζόμενοι, αλλά τα κράτη-μέλη ή οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να το μειώσουν. Το μόνο σημείο που πρέπει να διευκριστεί ακόμη για το πεδίο εφαρμογή είναι ότι η έκθεσή μου δεν έλεγε τίποτα για την ε, ιδιαίτερη πραγματικότητα για τις αναδιαρθρώσεις που δεν, αφορά μόνο, δεν αφορούν μόνο τον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε μέσω αυτής της οδηγίας να ασχοληθούμε με τον στενό δημόσιο τομέα. Αλλά αυτό που κάνω στην ε, τροπολογία 119 είναι να λέω ότι στο δημόσιο τομέα υπάρχουν ε, ε, εταιρείε, υπάρχουν επιχειρήσεις με εμπορικέ δραστηριότητες και θα μπορούσαν λοιπόν να συμπεριληφθούν. Το δεύτερο πρόβλημα που έθεσαν οι εμπειρογνώμονες είναι ότι επειδή είναι περίπλοκο πολύ το θέμα αυτό υπάρχουν ε, πολλές οδηγίες που ήδη, ναι, ναι, τελειώνω, πολλές οδηγίες που απασχολούνται με, που ασχολούνται με διάφορους, ε, διάφορα τμήματα του τομέα αυτού. Αυτό ε, τα συνδικάτα κυρίως τονίζουν είναι ότι αυτές οι οδηγίες ε, καλύπτουν με μεμονωμένους τομείς αλλά δίνουν κάποιες εγγύσεις για ενημέρωση κτλ. Και, ότι με αυτή την ενιαία τώρα οδηγία μπορεί να θίγονται αυτές οι εγγύσεις για την ενημέρωση και άλλες δυνατότητες συμμετοχής των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν με τη δική μου τροπολογία τονίζω στην 155 τονίζω ότι πρέπει να γίνεται διαβούλευση για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και αναφέρομαι και στην νομοθεσία για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και για τα συμβούλια εργαζομένων και με άλλη τροπολογία μου λέω ότι πέρα από τα θέματα που, υπάρχει, που αναφέρονται στην οδηγία μου υπάρχει και εθνική νομοθεσία για την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους και συνολικότερα. Τρίτο θέμα. Τα συνδικάτα ανησυχούν ιδιαίτερα για το ότι επειδή θέτουμε ελάχιστε προδιαγραφέ, ίσω να μην ήταν δυνατόν να βελτιωθούν. Εγώ βάζω μια ρήτρα εδώ, που είναι πολύ χαρακτηριστική σε όλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ότι αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα, τη δυνατότητα των κρατών να υιοθετήσουν πιο ευνοϊκά μέτρα. Δύο θέματα, κυρία Πρόεδρε. Σημαντικά. Η πρώτη είναι η ανησυχία για το σεβασμό των εθνικών νομοθεσιών και των συλλογικών συμβάσεων. Όλες οι υποχρεώσεις, αυτό το λέω στην τροπολογία 47 με μια νέα αιτιολογική σκέψη, λέμε με μεγάλη σαφήνεια, ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμός όλων αυτών. Εμείς είμαστε ελάχιστες προδιαγραφέ που εφαρμόζεται μόνο όταν δεν υπάρχει καθόλου κοινωνική προστασία ου μέσω συμβάσεων. Στην 152 τροπολογία το ίδιο θέμα καθορίζουμε ότι η αναδιάρθρωση είναι αυτή που ορίζει ο εθνικός νόμος για να μην υπάρχει καμία απόκληση. Στην τροπολογία 18 αναφέρω κάτι που μου ζητήθηκε επίσης και που νομίζω ότι είναι κατάλληλο. Γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα ούτε για το εθνικό δίκαιο, για τις συλλογικές συμβάσεις, ούτε για τις επιχειρήσεις. Μόνο αυτό που είναι απόλυτα ε, κατάλληλο. Και σε άλλες τροπολογίες λέω τα ίδια, γιατί κάποια κρατημένη, κάποιες μόνιμες αντιπροσωπείες επέμειναν ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η εθνική νομοθεσία που ήδη υπάρχει για τη χρήση βιομηχανικών ζωνών ε, που είναι πια απερχιωμένες. Βεβαίως, βεβαίως. Θα σεβαστούμε, όπως λέει η 312, την άποψη των κρατών μελών για τις βιομηχανικές περιοχές και η εμπιστευτικότητα. Βεβαίως. Θα γίνεται με βάση τους ε, εθνικούς ορισμούς για την ε, εμπιστευτικότητα. Δεν υπάρχει μόνο μία λοιπόν εμπιστευτικότητα. Τα κράτη-μέλη, κατά λίγο, κατά λέγοντας ότι υπάρχουν και άλλε τέσσερι τροπολογίε. που είναι στο πνεύμα αυτών που επιχειρώ να κάνω. Είναι τροπολογίες που προσπαθούν να επιτύχουν ισορροπία με βάση αυτά που έλεγε και ο πρόεδρος της Business Europe. Θέλουμε να υπάρχει ελαστικότητα αλλά και ασφάλεια. Ελαστικό ασφάλεια. Θέλουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ελαστικότητα από μια μεριά και την ασφάλεια που απαιτούν εργαζόμενοι. Εδώ είναι η ουσία της υπόθεσης. Προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία μεταξύ ελαστικότητας και ασφάλειας. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να απορριφθεί. Για τις αναδιαρθρώσεις λοιπόν προτείνω στην τροπολογία 84 οι επιχειρήσεις για να καταλάβουν δηλαδή ότι δεν είμαι κατά των επιχειρήσεων, είναι κάτι που πρότεινε επιχειρήσει. Οι αναδιαρθρώσεις τι καθορίζω σαφώς, Που επιδιώκουν τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα. Καταλαβαίνω ότι χρειάζονται κάποια ελαστικότητα επιχειρήσει. Αλλά παράλληλα το αντιστάθμισμα είναι να καταλάβουμε ότι οι εργαζόμενοι που κάνουν τη δουλειά του να έχουν δικαίωμα για μια κατάρτιση, σε βοήθειε, αν και βέβαια οι εργαζόμενοι, όπω λέω στην τροπολογία 93, θα, έχουν, θα πρέπει να αναλάβουν την υποχρέωση να ε, εκπαιδευτούν εκ νέου. Σίγουρα είναι πολύ χαρούμενοι όταν του δίνουν τέτοιε δυνατότητε. Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση των επιχειρήσεων να του προσφέρουν και υποχρέωση των εργαζομένων να δεχτούν την επανεκπαίδευση. Η ελαστικό ασφάλεια σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Και οι τροπολογίε που πρότειναν τα συνδικάτα το καθορίζουν αυτό. Κάτι που με πρότεινε το Δουβλίνο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε σύστημα ενημέρωση ε, καλό για τι αναδιαρθρώσει. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι, διακόπτη πρόεδρο, οι εργαζόμενοι δουλεύουν με βάση άρθρα στον τύπο. Καταλήγω λέγοντα ότι η τελευταία τροπολογία προσπαθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε ένα σύστημα ενημέρωση που να μα επιτρέπει να εργαστούμε στο μέλλον. Ελπίζω την επόμενη φορά να ζητήσουμε αναλυτικά ένα θέμα που δυστυχώ πρέπει να αντιμετωπίζουμε, αλλά που νομίζω ότι είναι στην μέση διάταξη εκατομμύρια εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό να τα πούμε όλα αυτά και είναι σημαντικό και οι υπόλοιποι να μπορέσουν να πάρουν το λόγο και μας μένουν πέντε λεπτά μόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μπω στην ουσία των τροπολογιών. Είναι πρόωρο νομίζω πρέπει να συναντηθούμε ούτως ώστε, όπως είπε και ο, ο κύριος Θέρκας, επειδή είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, πολύ σημαντικό το θέμα, οπότε πιστεύω ότι είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναβλήθηκε η ψηφοφορία και που έχουμε λοιπόν μέχρι τον Νοέμβριο για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι για όλους μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Όλοι θέλουμε να υπερασπιστούμε και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να συνεχίζουν να μεταφέρονται αυτές οι επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε το αναγκαίο, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε συνενέσεις. Υπάρχουν κάποιε αμφιβολίε, είναι σαφές, για το εάν και κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να προκρίνουμε οδηγία ή άλλο είδος. Μπορούμε πιστεύω να... ότι πρέπει να επιχειρήσουμε να καταλήξουμε σε μια νομική μορφή που να είναι πάνω από σύσταση αλλά να μπορεί να αποτελεί αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας και για αυτούς που δεν θέλουν οδηγία. Πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές για όλες τις χώρες. Αλλά επίσης αναμφίβολα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε αυτό. Γιατί σε κάθε κράτος υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές, διαφορετικά πρότυπα. Πρέπει να επιδιώξουμε να καταλήξουμε στους ίδιους κανόνες ή κάποιους ελάχιστους κανόνες που να ισχύουν για όλους. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, θα εργαστούμε πολύ και ως εκπρόσωπος ε, του ΕΛΚ για το θέμα αυτό ελπίζω να καταλήξουμε σε συνένεση. Μπορείτε να βασιστείτε στη συνεργασία μας για να καταλήξουμε λοιπόν σε συμφωνία για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Είμαι στη διάθεσή σα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με όλους τους άλλους για να επιδιώξουμε ε, συνένεση που νομίζω ότι είναι σημαντική. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη δουλειά σας. Ξέρω με πόσο μεγάλη ένταση και προσπάθεια επιτελείται το έργο του εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καζίνη και μετά Κορνέλισεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορεί κανείς παρά να σεβαστεί τις προθέσεις του εισηγητή. Τα κίνητά του είναι μια ξεκάθαρη άποψη, έτσι ώστε οι αναδιαρθρώσεις να είναι όσο λιγότερο δίνει ρες γίνεται, αλλά δεν συμμεριζόμεθα τους στόχους, συμμεριζόμεθα τους στόχους μεν όχι όμως και τα μέσα. Έχουμε διαφορές για τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τις επιχειρήσεις και τις αναδιαρθρώσεις. Οι επιχειρήσεις και οι αναδιαρθρώσεις δεν είναι κάτι κακό που πρέπει να αποφευχθεί, αλλά είναι μια επιχειρηματική, επιθυμητή συχνά διαδικασία που θα καταστήσει πιο κερδοφόρες τις επιχειρήσεις και θα τις προσαρμόσει καλύτερα στις οικονομικές συγκυρίες. Γι' αυτό ακριβώς δεν φαίνεται στην έκθεση ότι οι επιχειρήσεις είναι κάτι το δεδομένο. Πολλές παράγραφοι ζητούν από επιχειρήσεις προφανή μέτρα, τα οποία έτσι και αλλιώς προς το συμφέρον τους μακροπρόθεσμα πρέπει να εφαρμόσουν, αλλά κάτω από συνθήκες κρίσης κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αντισκαταστρέψει βραχυπρόθεσμα λόγω των εξαιρετικών ποσοστών, υψηλών ποσοστών ανεργίας σε πολλές χώρες. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο μπροστά μας τις θέσεις απασχόλησης ποιοτικέ και μακροπρόθεσμες. Εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν κάθε είδους εργασία και δεν είναι σε θέση να είναι επιλεκτικοί, όπως ούτε και εμείς. Τελικά, μόνο μια επικερδής εταιρεία θα μπορέσει να διασφαλίσει θα έλεγα μια δυνατότητα επιβίωσης χωρίς απώλεια θέσεων απασχόλησης. Μόνο με ένα σωστό ισολογισμό θα μπορέσει να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους έτσι ώστε να παραμείνουν χρήσιμοι στο μέλλον. Απαιτείται μια πιο ευέλικτη διαδικασία και έτσι πολλές από τις συστάσεις τις οποίες κάνουμε εμείς στην έκθεσή μας θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν καθοδηγητήριες γραμμές θα έλεγα και παραδείγματα βέλτισης πρακτικής. Θα υποστηρίξουμε κάθε λογικό μέτρο για την προστασία των εργαζομένων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προετοιμάσουν και τους εργαζομένους τους όπως είπατε. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε όμως να εξισορροπήσουμε τα μέτρα αυτά έτσι ώστε να μην τα καταστήσουμε ένα επιπλέον βάρος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, θα έλεγα μια απώλεια την οποία δεν μπορούμε να υποστούμε πλέον. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι παρά τις διαφωνίες μας θα είμαστε ανοιχτοί σε επικοδομητικό διάλογο με όλους. Το χρονοδιάγραμμά σας το αποδεχόμεθα διότι μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Κυρία Κορνέλησεν, ευχαριστώ τον κύριο Κατσίνη. Έχω απογοητευτεί λίγο από τη στάση των φιλελευθέρων απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, ομολογώ. Το να λέμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε επιλεκτικοί σε σχέση με τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και αν είναι αξιοπρεπείς οι θέσεις αυτές είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ξεχωρίζει μια αξιοπρεπή επιχείρηση από τις υπόλοιπες. Οι θέσει απασχόλησης πάντα πρέπει να είναι αξιοπρεπείς. Και αυτό που είπατε για λογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων είναι θέμα ορισμού, δεν ξέρω τι εννοείται. Πάντως θα δούμε αν μπορούμε στα πλαίσια των συμβιβαστικών προσπαθειών να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία. Εκεί που θα συμφωνήσω είναι ότι η αναδιάρθρωση από μόνη της δεν είναι κάτι το αρνητικό στα πλαίσια μιας δυναμικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιδρούν δυναμικά. Και αν θέλουμε να υπάρξει μετάβαση και στην πράσινη οικονομία όπως όλοι το επιθυμούμε, τότε οι αναδιαρθρώσεις είναι απαραίτητες και αναπόφευκτες. Απαιτούνται όμως κάποια ελάχιστα επίπεδα σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τη μεταχείριση των εργαζομένων τους. Υπάρχουν τόσο αποκλίνουσες πρακτικές στα διάφορα κράτη-μέλη. Σε ορισμένες χώρες απαιτούνται να υπάρχουν σαν παράδειγμα κοινωνικά προγράμματα, να δίδονται επιδοτήσεις για κοινωνικούς λόγους, να επανεκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι αν είναι αυτό απαραίτητο, ενώ σε άλλες χώρους σε άλλε χώρε, συγγνώμη, πρέπει να ενημερώνει του εργαζομένους μόνο και μόνο μοναδική υποχρέωση έξι εβδομάδες πριν. Λοιπόν, υπάρχουν πολλέ διαφορέ και χρησιμοποιούνται και οι εργαζόμενοι και η ασφάλειά του πολλέ φορέ για ανταγωνιστικού λόγου και στα πλαίσια του EGF η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλέ φορέ καλείται να πληρώσει το λογαριασμό για εταιρείε σε χώρε στις οποίε δεν υπάρχουν καθόλου κανόνε ενώ σε άλλε χώρε. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες οφείλουν να πληρώσουν το κόστος. Σύμφωνο λοιπόν με την έκθεση του κυρίου Σέρκας, με την πρώτη προσπάθειά του να καταλήξουμε σε κοινά ελάχιστα επίπεδα προστασίας, θα θέλαμε σε ορισμένους τομείς να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά είναι απαραίτητο να δούμε και το τι είναι πολιτικά εφικτό πλέον. Από ό,τι καταλαβαίνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τώρα που της πετάξαμε την μπάλα θα κάνει τις δικές της προτάσεις. Φυσικά θα υπάρξει μέχρι τότε μια πολιτική και ιδεολογική μάχη μέχρι τη στιγμή της κατάθεσης της τελικής πρότασης και θα πρέπει να πετύχουμε την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία και να συνεχίσουμε τη συζήτηση και με τον κύριο Κασίν, έστω και στους διαδρόμους, για να τον πείσουμε. Κύριε Θέρκας, δεν έχουμε άλλο χρόνο για τη διαμηνία. Έχετε ένα λεπτό μόνο για να κλείσετε τη συζήτηση. Ένα λεπτό για να ευχαριστήσω τις ε, προσφορές διαλόγου. Δεν θα πέσουν σε άγωνο έδαφος. Θα ήθελα ε, να πω στη φίλη Βερόνικα, στον κύριο Κασίν, σε όλους που πήραν το λόγο, ε, να τους πω αυτό που πριν από μια εβδομάδα είπα στον κύριο Μπαρόσο. Του είπα ότι η παγκοσμιοποίηση απαιτεί ενιαία απάντηση και την απάντηση αυτή δεν θα την καθορίσουν οι πιο βραδιπορούντες. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη κοινωνική Ευρώπη. Ο κ. Φερχόφστατ μίλησε για μια Ευρώπη ως συνομοσπονδία πολιτών. Ελπίζω λοιπόν ότι ένα τέτοιο θέμα που ε, από το οποίο έχουν τεράστιες προσδοκίες οι πολίτες όταν μιλάμε για ένα συμβόλαιο με τους ε, πολίτες, βεβαίως, βεβαίως όλα τα νόμιμα συμφέροντα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όχι και στο μέλλον δεν θα είμαστε καθυστερημένοι, αλλά πρέπει να κάνουμε ζωμένα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα άλλο. Je disais donc Έλεγα λοιπόν ότι επί τη βάση αυτή της ενεργού ε, συνεργασίας στι 9 Οκτωβρίου θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων ε, για τη μονάδα που ασχολείται με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του Κοινοβουλίου. Θα είναι η πρώτη φορά και μάλλον θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα εξετάσουμε ταυτόχρονα ε, τις τροπολογίες. Φαντάζομαι ότι μέχρι τότε θα έχουμε συμβαστικές τροπολογίες, τόσο να εγκριθούν σε έκτακτη συνεδρία στις 5 ή τις 6 Νοεμβρίου. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας ε, για το πρωί. Σας προσκαλώ όμως ε, ε, για να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Ποζίτσα που πλέει προς νέα και ενδιαφέροντα πελάγη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελάτε λοιπόν ε, αν θέλετε σε ένα κοκτέιλ που θα γίνει ε, έξω από την αίθουσα. Ευχαριστώ.